Ξεκινάμε τη συνεδρίαση, λέει ο Πρόεδρος. Ας εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Αλλά να σας πω και κάποια πράγματα. Έχουμε μια-δύο μικρές αλλαγές στην ημερήσια διάταξη. Η έκθεση Γκάιερ, το σημείο 15, για την απαλλαγή 2009, ζητήθηκε να ψηφιστεί τελευταίο διότι δεν μπορεί να παρίσταται, έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις. Φορέστε τα ακουστικά σας για να μ' ακούτε. Σας είπα λοιπόν συνάδελφοι ότι αλλάζουμε την ημερήσια διάταξη. Ο κύριος Γκάιερ που τον έχουν στο σημείο 15 παρακάλεσε η έκθεσή του να ψηφιστεί τελευταία στο κατάλογο λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων που σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι εδώ τώρα. Και άλλη μια αλλαγή. Ανταλλάσσουμε τα σημεία 10 και 11. Διότι η κυρία Μπαλτσάνη, η Γενική Συγκίτρια για τον Προπολογισμό 2012, το ζήτησε. Να έρθει στις 9.30. Λοιπόν, αν συμφωνείτε με αυτές τις δύο αλλαγές, μπορούμε να θεωρήσουμε ως εγκεκριμένη την ημερήσια διάταξη. Δεν βλέπω σχόλια. Άρα εγκρίνεται η μερίσια διατάξη. Ω συνήθως, η συνεδρίασή μας εκπέμπεται στο διαδίκτυο μέσω web streaming. Πάμε στο σημείο 2 της ημερήσια διάταξη, Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 14 η και τη 28 η Φεβρουαρίου. Θεωρούνται συγκεκριμένα τα πρακτικά, εφόσον βλέπω ότι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, ή αν δεν ακούσουν κατά τη διάρκεια τη συνεδριά σα. Πάμε στο σημείο 3. Έχω να σα ενημ... πω κάποια πράγματα. Ότι οι συντονιστέ θα πάρουν αποφάσει και θα σα ενημερώσω αύριο σχετικά με αυτέ. Την περασμένη εβδομάδα, το 16 Μαρτίου, συμμετείχαμε στη δεύτερη συνάντηση της Task Force Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Αμοιβαιότητα και είχαμε το μνημόνιο συνεννόηση από την πρώτη συνεδρίαση και πληροφορίες επίσης σχετικά με τη δεύτερη συνεδρίαση θα σας διανεμηθούν. Πάμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Έκθεση του Μάικλ Τόρερ που αφορά την απορρόφηση των πόρων των διαθροτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, συναγόμενα διδάγματα για την πολιτική συνοχή της Ένωσης και θα παρακαλούσα τον εισηγητή να κάνει με σύντομη εισαγωγή. Θα έχουμε περίπου μισή ώρα για την συζήτηση. Ναι, αγαπητοί κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η παρθενική μου έκθεση για ένα θέμα το οποίο σας ενδιαφέρει όλους. Τα θέματα των ποσοστών απορρόφησης και τα προβλήματα απορρόφησης των διαρθρωτικών ταμείων για το Ταμείο Συνοχής. Στο παρελθόν έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις για τα θέματα αυτά και έχω τώρα φτάσει στο σημείο της διατύπωσης ενός εγγράφου εργασίας. Προφανώς δεν είναι η οριστική έκθεση. Περιλαμβάνει μερικές βασικές ιδέες οι οποίες θα πρέπει να κατευθύνουν τη συζήτηση και προφανώς το θέμα αυτό της ε, απορρόφησης των, του Ταμείου Συνοχής είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία έχουμε συζητήσει πολλές φορές και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά έχει προκαλέσει και συζητήσεις και στα κράτη-μέλη και στις περιφέρειες της Ευρώπης με τόσα πολλά λειτουργικά προγράμματα δεν είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς ποιο είναι το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων. Γενικά όμως έχουμε προβλήματα. Ο στόχος μας λοιπόν θα πρέπει να είναι να συλλέξουμε στοιχεία και να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες για το πού βρίσκονται τα προβλήματα και αν υπάρχουν κάποια γενικά σχήματα τα οποία να είναι παρόμοια στις περιοχές όπου στις όπου εφαρμόζονται αυτά τα κονδύλια, ώστε να μπορέσουμε να αντλήσουμε κάποια συμπεράσματα γενικού χαρακτήρα. Αλλά για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο χρειαζόμαστε καταρχήν μια βάση πληροφόρησης, μια βάση στοιχείων. Και ο στόχος μας είναι να συζητήσουμε με την Κομισιόν πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη συλλογή αυτών των στοιχείων για να έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία μας είναι απαραίτητα Όπω ξέρετε, στι εισηγμένε στο χρηματιστήριο εταιρείε ζητάμε τριμηνιαίες εκθέσεις. Δεν θα ήταν παράλογο λοιπόν να έχουμε και τριμηνιαίες εκθέσεις για τα λειτουργικά προγράμματα στο Ταμείο Συνοχής, αλλά αυτό δεν είναι ο μόνος τρόπος. Το ζήτημα είναι να ξέρουμε πώς ε, μπορούν μπορεί το Κοινοβούλιο να γνωρίζει για, την, για τα κονδύλια και την απορρόφησή τους, ώστε με τον τρόπο αυτό να έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε με την Κομισιόν και με τα κράτη-μέλη για το πώς να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα τα οποία αναφύονται. Είναι λοιπόν η έκθεση αυτή μια γενική επισκόπηση στον τομέα αυτό, καταδεικνύει ποια είναι τα προβλήματα, αλλά αναφέρεται και στις βέλτιες πρακτικές για την τρέχουσα περίοδο 2007-2013 και θα πρέπει να τροφοδοτήσει και την περαιτέρω συζήτηση και θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου με, για την συνεργασία που είχα από τους σκιώδεις εισηγητές των άλλων πολιτικών ομάδων <clears throat> οι οποίοι μου έχουν παρουσιάσει τις απόψεις τους για τα συμπεράσματα τα οποία μπορούμε να αποκομίσουμε από τη μελέτη της απορρόφησης των ταμείων αυτών και έχουμε και δύο ουσιαστικά την επικάλυψη δύο περιόδων ε, προγραμματισμού επικαλύπτεται σε κάποιο βαθμό η περίοδος 2000 με 2006 και 2007 με 2013 σε ό,τι αφορά την ε, χρηματοδότηση και την ε, εκταμείευση των κονδυλίων γιατί ξεκινήσαμε αρκετά αργά με την εφαρμογή ορισμένων λειτουργικών προϊόντων επειδή υπήρχε μία ασάφεια σε σχέση με την χρηματοδότηση και αυτό οδήγησε και συζητήσει σε σχέση με τους κανόνες νησιν 2 και νησιν 3. Επίσης, η παγκόσμια ύφεση οδήγησε σε μεγάλα προβλήματα στα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την συγχρηματοδότηση. Επιπλέον υπήρξαν και περαιτέρω κανονιστικές απαιτήσει και ρυθμίσεις για διαορισμένε περιοχές. Αναφέρονται επίσης προβλήματα συμβατότητος, ιδιαίτερα ιδιαίτερα σε ορισμένα κράτη-μέλη, τα οποία ακολουθούν εθνικούς κανόνες οι οποίοι δεν συνάδουν πάντα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες ή ορισμένε φορές βρίσκονται σε σύγκρουση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και επομένως πρέπει να υπάρξει κάποια διαλεύκανση αυτών των κανόνων. Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη να ευθυγραμμίσουμε καλύτερα τους εθνικούς κανόνες με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξάλλου διαπιστώσαμε ότι υπάρχει και ασάφεια σε ορισμένε περιοχέ, υπάρχουν κενά στην νομοθεσία σε ορισμένα κράτη-μέλη σε σχέση με του κανόνε που πρέπει να εφαρμοστούν. Επίση, υπήρξαν και προβλήματα για τη λήψη απόφαση σε ορισμένα κράτη-μέλη σε σχέση με την ε, ιεραρχία Λήψη απόφασης και υπήρξαν και ανεπαρκείς ε, μορφές διαχωρισμού μεταξύ των αρμοδίων αρχών και πολλές φορές υπήρξαν πολλαπλοί φορείς οι οποίοι έπρεπε να εξετάσουν τα ίδια θέματα, κάτι το οποίο δυσκολεύει τη διαδικασία. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε επίσης και προβλήματα ικανότητας εφαρμογής σε περιφερειακό επίπεδο, ακόμα και σε εθνικό επίπεδο σε ορισμένε περιπτώσει, που θα πρέπει να βελτιωθεί αυτή η ικανότητα υπήρξαν προβλήματα παραγωγικά με τη μηχανογράφηση, τα συστήματα τεχνολογίας πληροφορία και την εφαρμογή των εθνικών κατευθυντηριών γραμμών. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα αυξημένος έλεγχος για τα προγράμματα αυτά και τις χρηματοδοτήσεις. Το ερώτημα είναι αν αυτό θα οδηγήσει και σε περισσότερες ε, συγκρούσεις, δηλαδή η ο μεγαλύτερος έλεγχος αν θα οδηγήσει σε προβλήματα για την απορρόφηση σε περαιτέρω προβλήματα. Το ερώτημα είναι πώς θα μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη απορρόφηση αλλά συγχρόνω και καλύτερο έλεγχο. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι χρήσιμο και πρόσφορο να σκεφτούμε αν μπορούμε να βρούμε τρόπους απλοποίησης των διαδικασιών ώστε να έχουμε μεγαλύτερη αποδοτικότητα και να αποφεύγουμε τα σφάλματα. Θα έπρεπε να σκεφτούμε λοιπόν καλύτερα αν θα πρέπει η αστίαση να είναι στον έλεγχο του προπολογισμού και την ε, επαγρύπνηση για, το, για να μην υπάρξουν ατασταλίες και απάτες και αν θα πρέπει να δώσουμε εδώ πέρα μεγαλύτερη έμφαση στην τυπική εκπλήρωση όλων των κανόνων. Πρέπει όμως να εξασφαλίσουμε και μια μεγαλύτερη αναλογικότητα μεταξύ του μεγέθους των κονδυλίων και της επάχθειας του ελέγχου. Και εδώ πιστεύω το, το σύνθημα η βασική ιδέα είναι ότι δεν θα πρέπει για ψηλά, για θέματα τα οποία είναι πραγματικά πενταροδεκάρες, να εφαρμόζονται πολύ βαριοί κανόνες ελέγχου. Είναι μεγάλη σημασία επίσης να εξασφαλίσουμε ότι και στο μέλλον θα είμαστε σε θέση να εξασφαλίσουμε μια χρηματοδότηση για το Ταμείο Συνοχής μέσα στις επερχόμενες δημοσιονομικές προοπτικές και εξάλλου τονίζω και πάλι την ανάγκη να υπάρξει καλύτερη αποδοτικότητα και εφαρμογή των διαθωτικών ταμείων. Δεν κάνω φυσικά μια εξαντλητική απαρίθμηση περιπτώσεων, απλώς δίνω κάποια παραδείγματα τα οποία περιλαμβάνουν ορισμένες σκέψεις σε σχέση με περιπτώσεις σε διάφορες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να τις σκεφτούν και τα κρατημέλη και το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό θα πρέπει να εμπλακεί σε αυτή τη συζήτηση και θέλω να σας υπογραμμίσω ότι η σημερινή συζήτηση είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψε με τα θέματα αυτά και εγώ χαίρομαι ήδη εκ των προτέρων για τις προτάσεις που μπορούν να προέλθουν από τους συναδέλφου και από τις υπόλοιπε πολιτικές ομάδες και εξάλλου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την, την, ε, ε, την ευκαιρία να ακούσουμε την άποψη της Επιτρόπης των Περιφερειών που έχουν μια πολύ καλή σύνδεση με τις περιφέρειες και την τοπική αυτοδιοίκηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένω, από όλε αυτέ τι πηγέ είμαι έτοιμο να δεχτώ προτάσει και φυσικά είμαι έτοιμο να ακούσω και αυτά τα οποία θα θελήσει να μα πει η Κομισιόν και το Συμβούλιο. Θέλω λοιπόν εκ των προτέρων να σα ευχαριστήσω για την συμμετοχή σας και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και τη γραμματεία της Επιτροπής που με βοήθησε ιδιαίτερα στην εκπόνηση αυτού του εγγράφου. Ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως είπε ο συγγετής, αυτό είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Θα εξεταστεί το σχέδιο εκθέσεω το Μάιο. Α ξεχνούμε του σκιώδεις Ο Βίκτορ Μποστινάρου θα πάρει το λόγο. Okay. Imagine that my colleague... Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι η Σοφία Κόν δεν είναι η Σοφή, Τέλο πάντων, έλεγα ότι ήθελα να μιλήσω ο συνάδελφο. Καλωσορίζω τι κατευθυντήριε γραμμέ που εισάγονται του συγκεκριμένου συνάδελφό μα, τον Μιχαήλ ε, Τόρερ, και να πω, χωρί να επεκταθώ, ότι κατά την άποψή μου αυτή η έκθεση δεν έρχεται μόνο έγκαιρα αλλά είναι και πολύ σημαντική διότι αφορά τη συζήτηση του μελλοντικού δημοσιονομικού πλαισίου. Είναι πολύ σημαντικό να αντλήσουμε τα μαθήματα από το παρελθόν για να βελτιώσουμε το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Πρέπει να βρούμε τρόπο να αυξήσουμε τη δυνατότητα απορρόφησης σε αυτό το εργαλείο. Βλέποντας τα αριθμητικά στοιχεία, Υπάρχουν ανησυχητικά αριθμητικά στοιχεία εντό τη εκθέσεω και εντό των προσανατολισμών που παρουσιάζει σήμερα διακεκριμένο συνάδελφο, ο κ. Τόιραρ. Καταρχά, να σα πω ότι είναι ζωτική σημασία στο μέλλον να συζητήσουμε ποια μέτρα μπορούμε να εφαρμόσουμε για να αυξήσουμε το διοικητικό δυναμικό. Και επίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει στο μέλλον στι συμβάσει για αναπτυξιακή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 100 μελών να συμπεριλαμβάνει στοιχεία συγκεκριμένα που καμιά φορά θα είναι δεσμευτικά, ούτω ώστε να πιέζονται τα κράτη-μέλη και έτσι να συμμορφώνονται πλήρω, λαμβάνοντα τα αναγκαία μέτρα με τι επιταγέ του πλαισίου και να αποφύγουμε τη σημερινή κατάσταση στο μέλλον. Δύο, Η δυνατότητα απορρόφηση. Αυτό αφορά και εκείνους που εργάζονται στη δημόσια δίκηση των κρατών μελών. Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε ένα θεσμικό πλαίσιο για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα και που ασχολούνται με την ε, υλοποίηση των μέτρων αυτών τη Ευρωπαϊκή Ενώση. Πρώτα απ' όλα σταθερότητα. Πρέπει να υπάρχει σταθερότητα όσον αφορά του εργαζομένου που ασχολούνται με την απορρόφηση και το δυναμικό απορρόφηση. Δεύτερον, να δώσουμε κίνητρα. Να πληρώνονται καλά αυτοί οι άνθρωποι, ούτω ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά του. Να είναι αποτελεσματικοί. Στη Ρουμανία, όπου πληρώνονται πολύ λίγο οι υπάλληλοι και δεν έχουν κανένα κίνητρο, να εργαστούν για την απορρόφηση εκατομμυρίων. Είναι τοπικό να θεωρήσει κανείς ότι κάποιος που πληρώνει 200, πληρώνεται 250 ευρώ το μήνα θα κάνει εντυπωσιακή δουλειά όσον αφορά την απορρόφηση εκατομμυρίων. Διότι αυτό δεν μπορεί να σταθεί. Αυτό μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βελτιώσουμε αυτό το στοιχείο. Αυτό πρέπει να δούμε. Τρίτον, η πολιτική ανάμειξη, παρέμβαση, πώς θα αποφευθεί. Μπορεί να δηλωθεί ότι υπάρχει σταθερότης, αλλά θα πρέπει να αποφευθεί και πολιτική ανάμειξη σε θεσμικά όργανα που ασχολούνται με τη χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είναι κάτι που είναι γνωστό όχι μόνο στη Ρουμανία, αλλά και σε άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Είναι σημαντικό να υπάρχουν δεσμευτικοί κανόνες περί υποχρεώσεων. Υποχρεώσεων των κυβερνήσεων των κρατών μελών. Ποιε είναι οι υποχρεώσει σε επίπεδο περιφερειακών αρχών και ποια είναι τα δικαιώματα και υποχρεώσει σε επίπεδο τοπική αυτοδιοίκηση. Διότι ίσω να προσπαθεί η κεντρική κυβέρνηση να ελέγχει τα πάντα και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο είναι δυνατόν να μην έχουν λόγο οι τοπικοί φορεί. Και αυτό θα πρέπει να διορθωθεί. Η απλούστευση. Αναφέρθηκε σαφώ από τον κύριο Τόιλερ Ευπρόσδεκτη ιδέα. Και η Επιτροπή μας θέλει να το πετύχει αυτό. Είναι σημαντική συνεργασία με τους δικαιούχους όμως. Για να εντοπίσουμε σε μια κοινή προσπάθεια ποια είναι τα αναγκαία μέτρα. Τα μέτρα πρέπει να θεσπιστούν για να απλουστεύσουμε το σύστημα και να γίνει πιο προσβάσιμο. Εξακολουθεί να είναι περίπλοκο το σύστημα. Είναι ένα άχθος η γραφειοκρατία που βαρύνει τους ώμους της δημόσιας δίκησης. Άρα κάτι πρέπει να γίνει. Τέλος. Χωρίς να επεκταθώ, θέλω να πω το εξής. Είναι σημαντικό να υποβάλουμε τροπολογίες όταν θα έχουμε στα χέρια μας το σχέδιο κειμένου και στο τέλος είμαι σίγουρος ότι η Επιτροπή μας θα ετοιμάσει μία έκθεση που θα είναι επιτυχής, θα αποτελεί έμπνευση για μας, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τις μελλοντικέ μας συζητήσεις. Όταν θα έρθει η ώρα για να συζητήσουμε το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Βίκτορ. Ο Λάμπερτ Φαν Λίστερροϊ. Ευχαριστώ. Η κυρία είναι η σκιώδης εισηγήτρια, αλλά δεν έλαβε εγκύρα στο κείμενο. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και η κυρία Οκανή τον εισηγητή. Νομίζω ότι σωστά εντοπίσατε ε, το ότι συχνά επισημαίνονται στην αρχή της περίοδου της προγραμματικής δυσκολίες. Τώρα βρισκόμαστε στην ενδιάμεση φάση και θα μπορούσαμε να καταθέσουμε και κάποιες συστάσεις για τα χρηματοοικονομικά προβλήματα δώσαμε στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να έχουν συγχρηματοδότηση ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Μπορούμε να δούμε λίγο πιο πολύ σε βάθος γιατί σε κάποιες χώρες υπήρξε απορρόφηση και σε κάποιες άλλες όχι. Να μας πείτε επίσης τη γνώμη σας για τα άλλα οικονομικά μέσα. Το Τζέρεμι, τα νέα αυτά μέσα, τα οποία μπορεί να διδραματίσουν σημαντικό ρόλο να μην κοιτάμε δηλαδή μόνο προς τα πίσω, αλλά να δούμε και τι έχει γραφτεί στην πέμπτη έκθεση συνοχής και, και στην δική μας έκθεση. Και όντως ίσως θα πρέπει να κοιτάξουμε και τι γίνεται στις χώρες γιατί κάποιες ε, χώρες ε, όντω διπλασιάζουν τους διοικητικούς τους ελέγχους και αυτό εξαρτάται από την χώρα. Αν θα γίνει αυτό σε περιφερειακό επίπεδο, σε κρατικό επίπεδο, αυτό κατά πόσο επηρεάζει το αποτέλεσμα. Και επίσης, πολλές φορές το έχουμε συζητήσει. Έχουμε συζητήσει την περίπτωση κεντρικών ή μη κεντρικών ε, κρατών. Επηρεάζει αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει, για παράδειγμα, όταν θέλει κανείς να προσελκύσει επενδύσεις, να έχει σωστή ρύθμιση. Να σας πω ότι η κυρία Οκανή θέλει να τοποθετηθεί για το ενιαίο ελεγκτικό πρόγραμμα και τον έλεγχο που προβλέπετε. Επί του παρόντος, να σας πω ότι είναι πάρα πολύ έντονες οι κριτικές από τους συναδέλφους και η έκθεσή σας μπορεί να κάνει τη διαφορά, γιατί κάποιες χώρες θα πηγαίνουν εξαιρετικά, κάποιες χώρες θα πηγαίνουν χάλια. Και αυτές οι διαφορές σε μια τέτοια έκθεση καλό είναι να κατανομαστούν. Γιατί όχι. Θα μπορούσαμε να βάλουμε λίγο πιο πολιτικό χαρακτήρα, θεωρούμε εμείς. Uh, thank you. Ευχαριστώ. Βλάσακ. Ότζι paní Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θεωρώ ότι υπάρχει και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό από πλευρά των δικαιούχων. Να διασφαλιστεί ότι οι διάφοροι έλεγχοι θα έχουν μία συνέπεια, μία συνέχεια γιατί υπάρχουν κρατικοί έλεγχοι, τα σώματα τα εφαρμαστικά κάνουν τέτοιου ελέγχου. Και θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να γίνονται διάφοροι έλεγχοι για το ίδιο θέμα, αλλά να υπάρχει μια συνέχεια και να διαβιβάζονται οι πληροφορίε αυτές. Ούτε... Ο Ευγένη Κυρίλοφ είναι επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Τα προγράμματα της απορρόφησης είναι προβλήματα τα οποία υπάρχουν και συνεχίζουν να υπάρχουν. Είναι απαραίτητο να αναλύσουμε την κατάσταση αυτή και να δούμε ποια είναι τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν για το μέλλον. Εμείς δεν έχουμε συλλέξει στη χώρα μου όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να υπολογίσουμε το ποσοστό απορρόφησης και υπάρχει ίσως ε, μια διαφορά μεταξύ αυτών που έχουν δοθεί στους ε, τελικούς αποδέκτες και αυτών που έχει δώσει η Κομισιόν στη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία έχει, παραγωγός χάρη, 16% των κονδυλίων έχουν δοθεί στο κράτος και 11% στους τελικούς αποδέκτες. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των δύο αυτών στοιχείων. Είναι ανησυχητικά τα στοιχεία βέβαια αυτά. 22-23% είναι ο μέσος ρυθμός απορρόφησης, ενώ βρισκόμαστε στη μέση της περίοδου δημοσιονομικής σχεδίασης. Και υπάρχει και μία διαφορά μεταξύ των πρώτων στον κατάλογο και των τελευταίων στον κατάλογο. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν προβλήματα και ότι ορισμένα προβλήματα είναι πιο έντονα σε ορισμένες χώρες από ό,τι σε άλλα κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν να δούμε γιατί υπάρχει τόσο μικρό ε, ποσοστό απορρόφησης και γιατί είναι τόσο σημαντικά τα σφάλματα τα οποία έχουν διαπραχθεί. Είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε λοιπόν στο μέλλον την απλοποίηση των κανόνων και να, να καταλάβουμε τι είναι αυτά τα οποία μπορούν να διατηρηθούν στους ελέγχους και να ευνοήσουν ένα καλό ποσοστό απορρόφησης και ποια είναι τα στοιχεία ελέγχου τα οποία θα πρέπει να διαγραφούν. Και μπορούν τα κάτι μελη από μόνα τους να καθορίσουν δευτερογενείς κανόνες για τα θέματα αυτά. Θα ήταν χρήσιμο να δοθούν λοιπόν και ενδείξεις προς τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν μερικά κράτη τα οποία νιώθουν μεγάλη αγωνία γιατί φοβούνται ότι μπορεί να χρειαστεί να ε, δώσουν πίσω ορισμένα κονδύλια. Πολλές φορές κάνουν σφάλματα οι αποδέκτες γιατί δεν καταλαβαίνουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν για να δικαιολογήσουν τα κονδύλια αυτά. Τίθενται λοιπόν προβλήματα διοικητική ικανότητα και σε όλα τα επίπεδα και είναι απαραίτητο να προετοιμάσουμε σωστά όλα τα έγγραφα για, για τα επόμενα στάδια και να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να προετοιμαστούν για την επόμενη περίοδο δημοσιονομικών προοπτικών. Ούτε θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι δεν πρέπει να περιοριζόμαστε μονάχα στα αριθμητικά στοιχεία, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και το πραγματικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Euh, uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να συγχαρώ τον συνάδελφό μας για την πρωτοβουλία του. Αυτή η έκθεση κατά την άποψή μας ε, είναι ευπρόσδεκτη. Είναι φιλόδοξη έκθεση. Λαμβάνει υπόψη ότι είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί μια τέτοια ανάλυση αναλύση των λόγων για τους οποίους κάποια κράτη-μέλη είχαν καλή επίδοση και άλλα λιγότερο καλή. Μια τέτοια ανάλυση είναι περίπλοκη. Και σίγουρα χρειαζόμαστε μια τέτοια ανάλυση, κυρίως εν της επομένης προγραμματικής οικονομικής περίοδου, αλλά και για το χρόνο που μας απομένει θα τελειώσει η παρούσα περίοδος. Ελπίζουμε τα κράτη-μέλη που τώρα είναι σε πιο δύσκολη θέση να μπορέσουν να βρουν λύσεις για να βελτιώσουν το ποσοστό απορρόφησης πόρων. Αναφερθήκαμε στη γραφειοκρατία, στην αδυναμία του δημόσιου τομέα, στην ανεπάρκεια του δημόσιου τομέα, την έλλειψη ενθουσιασμού από πλευρά τη τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν έχει τόσο σημασία ο λόγο, πρέπει να βρούμε λύσει. Λύσει για να λύσουμε το πρόβλημα και για το τέλος αυτής της περίοδου προγραμματισμού, αλλά και για την επόμενη. Οι λύσεις, όπως η ενιαίοι έλεγχη, κοινοί κανόνες διαχείρισης των πόρων, των διαθωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, θα μπορούσαν να να αποτελέσουν λύσει. Έχουν δυναμικό. Ξανά τα συγχαρητήριά μου στον εισηγητή, τον κύριο Τόιρερ, και το εύχομαι καλή τύχη. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίο ομιλητή, Α, δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάτι να πει, να συμβάλλει στη συζήτηση. Ο Νίκολας Ματίν. Πρόεδρε, σα ευχαριστώ. Να απαντήσω στα σχόλια τα οποία ακούσαμε. Ασφαλώς, καταρχάς, ε, καλωσορίζουμε το ενδιαφέρον που επιδεικνύει η Επιτροπή σας για το θέμα αυτό και ασφαλώς το θέμα αυτό απασχολεί και εμάς και εσάς. Διαβάσαμε με προσοχή το σχέδιο της έκθεσης ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό και στις δικές μας τις σκέψεις για το θέμα αυτό, προφανώς. Εξετάσαμε την απορρόφηση κατά τα πρώτα έτη της προγραμματικής περίοδου για να δούμε ποιοι παράγοντες ε, θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν και για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Έχουμε λοιπόν πολλά στοιχεία τα οποία είναι κοινά με την δική σας έκθεση. Ένα επιπρόσθετο στοιχείο το οποίο θα θέλαμε να ρευτεί υπόψη και το οποίο δεν τονίστηκε ίσως αρκετά. Είναι η παράταση των προγραμμάτων για το 2000-2006. Πάντα υπάρχει μια επικάλυψη μεταξύ των ε, προγραμματικών περιόδων και ήταν ένα μέτρο το οποίο ε, το λάβαμε για να αντιποκριθούμε στην οικονομική κρίση. Να δώσουμε δηλαδή στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να επεκτείνουν, να παρατείνουν κατά έξι μήνες τα προγράμματα 2000-2006. Και αυτός είναι ένας από τους παράγοντες που οδήγησε και σε μια καθυστέρηση σε κάποια κράτη-μέλη προκειμένου να ξεκινήσουν τα καινούργια προγράμματα. Ένα γενικότερο σχόλιο που ήθελα να κάνω είναι ότι ασφαλώς το θέμα της απορρόφησης ήδη αντιμετωπίζεται στον κανονισμό με τον κανονα 1 NSYN2, 3 Αυτό είναι το πλαίσιο λοιπόν για να δοθεί ένα ισχυρό κίνητρο στα κράτη-μέλη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η απορρόφηση θα συνεχίσει με κάποια ταχύτητα. Γιατί το ξέρουμε ποιες θα είναι οι συνέπειες αν δεν ε, επιταχύνει η διαδικασία αυτή. Επίσης, ε, μία από τη συνέπεια της οικονομικής κρίσης ήταν να μεταρρυθμιστεί το NC2-NC3. Αυτή η μεταρρύθμιση τώρα θα αρχίσει να ισχύει. Αυτό θεωρώ ότι θα αποτελέσει ένα ισχυρό κίνητρο για τα κρατημέλη και επίσης κοιτώντας ε, ήδη την κατανάλωση των πιστώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2010 βλέπουμε ότι έχει αρχίσει μία πρόοδος. Αυτό φυσικά να πούμε ότι υπήρξε καλή απορρόφηση γιατί χρησιμοποιήθηκαν σε δικό μας επίπεδο στις δικές μας πιστώσεις 106% των προγραμμάτων. Αυτό είναι καλό λοιπόν, υπάρχει μια επιτάχυνση. Τώρα, για μια μέση τιμή χρήσης ε, των πιστώσεων για όλες τις χώρες και για το διευθυντικά ταμεία, 22%. Αλλά βλέπουμε όντως ότι υπάρχουν μεγάλες αποκλήσεις στα, στις χώρες ε, που υπήρξε καλή απορρόφηση. Είμαστε ήδη στο 30%. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα παθήματα που θα πρέπει να μας γίνουν μαθήματα, συμφωνούμε με αυτά που αναφέρονται στην έκθεση και υπάρχουν διάφορα στοιχεία, μερικά και των οποίων μπορούν να αντιμετωπιστούν με μελλοντικού κανονισμού. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη για να εναρμονιστούν όπου είναι δυνατόν αυτές οι καινούργιε νομοθεσίες. Και αυτό θα αφορούσε και την εναρμόνιση των ε, κριτηρίων ε, για τους ε, δικαιούχους. Αυτό είναι σημαντικό. Το έχουμε συζητήσει στο παρελθόν μαζί σας, θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να το συζητήσουμε. Επίσης συμφωνούμε ότι η διοικητική ικανότητα είναι εξαιρετικά σημαντική. Και το θέμα του να υπάρχει σταθερότητα μεταξύ των διαχειριστών των προγραμμάτων. Αυτή η άσκηση ποτέ δεν είναι εύκολη και απλή. Άρα είναι σημαντικό να διατηρείται η τεχνογνωσία και η εμπειρία που συλλαγεί κάθε άτομο μετά από κάποια χρόνια. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, το οποίο δεν είναι μόνο θέμα ρύθμισης, είναι να υπάρχει μία δίωδος για κάθε project. Εδώ επιμένουμε και θα επιμείνουμε και τα επόμενα χρόνια για να διασφαλίσουμε ότι όταν θα εγκριθούν τα καινούργια προγράμματα, οι αρχές διαχείρισης δεν θα αρχίσουν να ψάχνουν ε, project τα οποία θα πρέπει να συγχρηματοδοτηθούν, αλλά θα υπάρχει ένας καλός σχεδιασμός προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι δαπάνες επιτόπου. Άρα βλέπετε ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία. Δεν υπάρχει μία ενιαία μοναδική λύση. Υπάρχει μάλλον ένα συνδυασμό παραγόντων που επηρεάζει με διαφορετικό τρόπο κάθε χώρα. Και ασφαλώς θέλουμε να μάθουμε και από τις εμπειρίες του παρελθόντος σε ό,τι αφορά την νομοθετική διαδικασία. Αυτό θα το συζητήσουμε μαζί σας. Και για τα υπόλοιπα στοιχεία θα συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη προκειμένου να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τους κινδύνους που έχουμε εντοπίσει και τους οποίους και παρουσιάσαμε στην, στο σχέδιο έκθεσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Εξ ονόματος όλων των συναδέλφων να εκφράσω προς την Γενική Διεύθυνση Ρίζιο, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι περιμένουμε μία επίσημη αξιολόγηση της περίοδου 2007-2013 και της σχετικής απορρόφησης. Είτε φέτος, είτε στην αρχή του επόμενου έτους. Πότε θεωρείτε ότι θα μπορέσετε να μας δώσετε πιο αξιόπιστα στοιχεία μετά από ανάλυση σχετικά με την απορρόφηση. Και αυτό φυσικά θα μας πήγαινε λίγο παραπέρα από αυτό που συζητάμε σήμερα. Κυρία Πρόεδρε, τελειώνουμε τώρα την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το 2010. Κάναμε αρκετά λεπτομερή ανάλυση, συνεπώς, για να τιμάσουμε το κείμενο και να συναγάγουμε συμπεράσματα. Σίγουρα πριν το τέλος του Απριλίου θα είμαστε σε θέση να έρθουμε στην Επιτροπή και να σας παρουσιάσουμε τα βασικά στοιχεία της εκθέσεως και την ανάλυση του τι σημαίνουν αυτά τα στοιχεία όσον αφορά την απορρόφηση των πόρων μας στα διάφορα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Πολύ καλό, διότι θα ξανασυζητηθεί το σχέδιο εκθέσεως προς το τέλος Μαΐου. Οπότε και αυτή η συζήτηση ένα μήνα πριν θα είναι κάτι χρήσιμο για τον εισηγητή. Έχετε... Μάικαλ Τόρερ, έχεις το λόγο αν θες να πεις κάτι. Ναι, πολύ σημαντικό και περιμένω αυτή την ανάλυση διότι χρειάζεται πιο προσεκτική ανάλυση. Έχω δύο σχόλια. Αυτή η συζήτηση είναι η διαδικασία του άρθρου 50. Οπότε και η Επιτροπή επίσης συμπεριλαμβάνεται. Συμπεριλαμβάνεται και η ΙΜΚΟ. Οπότε θα μπορούσαμε να έχουμε ανταλλαγή μεταξύ συναδέλφων για να έχουμε μια κοινή θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν υπάρχουν αξεπέραστα εμπόδια. Δεύτερον, ενδιαφέρομαι για τη συλλογή παραδειγμάτων. Αν έχετε κάποια παραδείγματα με συγκεκριμένα προβλήματα, καλό θα ήταν να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ και προσλέπω στη συζήτηση. Πρόεδρος, ίσως να υπάρχουν και παραδείγματα πολύ καλής συμπεριφοράς, λέει ο Πρόεδρος. Δεν λαμβάνουμε απόφαση, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση τον Μάιο και ο εισηγητής κάλεσε εκείνους από εσά που θέλετε να συνεισφέρετε να ξεκινήσετε τώρα. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε για την ώρα των τροπολογιών. Ας πάμε στο σημείο 5. Η έκθεση του Γιάνν Αλμπριχτ για το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον ετήσιο προπολογισμό της Ένωσης. Θα ήθελα να προτείνω μια αλλαγή τη διαδικασία. Κανονικά ακούγεται πρώτα ο εισηγητή και παρεμβαίνει στο τέλο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχει αντίρρηση ο Γιάν. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με μια παρουσίαση τη δύσκολη από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μπορεί μετά εσύ να παρέμβει με σχόλια και ερωτήσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Νίκολα Μάρτιν εκ νέου. Από ό,τι καταλαβαίνω. Μπορείτε να κάνετε μια εισαγωγή, μπορείτε να μα εξηγήσετε τα βασικά στοιχεία και τα πιο δύσκολα γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολος αυτός ο κανονισμός. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω εν συντομία να εξηγήσω από πλευράς πολιτικής συνοχής ποιες θα είναι οι συνέπειες των προτινομένων αλλαγών στο δημοσιονομικό κανονισμό. Και αυτό σε σχέση με την όλη οργάνωση για την κοινή διαχείριση. Για να το κάνω αυτό, πρέπει εν συντομία να τονίσω ποιες είναι οι παρούσες ρυθμίσεις για έλεγχο, εποπτεία, δαπάνες για την πολιτική συνοχή για την περίοδο 2007-2013. Για να μπορέσω να σας παρουσιάσω και τα, τις αλλαγές που θα γίνουν από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τροποποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού. 2007-2013 λοιπόν. Έτσι που έχουμε σχεδιάσει το σύστημα για να ξέρουμε πώς θα πανώνται τα χρήματα ήταν να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται, πώς δημιουργείται το σύστημα ελέγχου μέσω της διαδικασίας αξιολογήσεως συμφο... συμμόρφωσης. Περιέγραψαν τα κράτη-μέλη το σύστημά του και μετά έγινε αξιολόγηση συμμόρφωση σε εθνικό επίπεδο. Εθνικό φορέα ελέγχου το έλεγξε και μετά τα πορίσματα επέλεξαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ εξέταση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά έδινε το πράσινο φω όταν ήταν ικανοποιημένη ότι όπω περιγραφόταν τα συστήματα συμμορφωνόταν με αυτά που θέλαμε. Αυτό κάναμε ευθύ εξ αρχή, από την αρχή τη περίοδου προγραμματισμού. Κατά τη διάρκεια τώρα τη υλοποίηση του προγράμματο υπήρχαν τρει βασικοί φορεί, τα κράτη-μέλη τα οποία ανεπλάκησαν στη διαχείριση των έλεγχο και την εποπτεία. Ο ελεκτικός φορέας χειρίζεται το πρόγραμμα και έχει πρωτίστως την ευθύνη για τον έλεγχο κατά πόσο είναι επιλέξιμα τα προγράμματα και κατά πόσο οι δαπάνε που παρουσιάζονται υπό συγχρηματοδότηση συμμορφώνονται με όλου του κανόνε και είναι νόμιμα μόνο με έξοδα και τακτικά, όπω πρέπει. Οπότε κάνει του ελέγχου πρώτο επίπεδο επιτόπου, στο επίπεδο του δικαιούχου. Μετά υπάρχει και ένας φορέας πιστοποίησης, είναι ένα δεύτερο ζευγάρι μάτια και εξασφαλίζει ότι οι δαπάνε είναι επιλέξιμες πριν αποσταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς ε, συγχρηματοδότηση. Κοιτάζει πάνω από τον νόμο του φορέα διαχείρισης, ούτως ώστε να διαπιστώσει ότι είναι καλή έλεγχη του φορέα ε, διαχείρισης και υπάρχει η διαβεβαίωση ότι οι δαπάνες πληρούν όλα τα κριτήρια πριν ε, δοθεί η αποζημίωση, η επιστροφή των χρημάτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάνει αυτή τη δουλειά η αρχή επιστοποίηση και επικυρώνει τι δαπάνε. Υπογράφει ένα κομμάτι χαρτί που λέει τα έλεγξα, όλα είναι καλά, όλα είναι νόμιμα, όπω πρέπει. Μπορείτε εσεί, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να πληρώσετε. Και ο τρίτο φορέα είναι ο ελεγκτικό φορέα, η ελεγκτική αρχή, εξωτερικό φορέα ελέγχου, ο οποίο ε, σαν έργο του έχει τον έλεγχο της σωστή λειτουργίας των συστημάτων. Έρχεται στο τέλο της διαδικασίας, εξετάζει τα συστήματα της αρχή πιστοποίηση και τη αρχής διαχείρισης, ούτω ώστε να είναι σίγουρος ο φορέας ότι λειτουργούν ομαλά και σωστά και για να δοκιμάσει αυτά τα συστήματα κάθε χρόνο ε, διενεργεί ελέγχους δειγματοληπτικά όσον αφορά τα διάφορα έργα και προγράμματα, ώστε να είναι σίγουρο ο φορέα ότι είναι επιλέξιμα όλα τα προγράμματα και νόμιμα. Είναι ένα τρόπο ελέγχου κατά πόσο οι έλεγχοι του πρώτου επίπεδου λειτουργούν ή όχι, εξετάζοντα ένα μικρό δείγμα όλων των επιχειρήσεων. Αυτοί είναι οι τρει βασικοί φορεί που υπάρχουν για την ώρα. Και από αυτή η πιστοποίηση από αυτή τη διαδικασία πηγαίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίω από την πιστοποίηση κάθε αξίωση πληρωμή και ετησίω μέσω γνωμοδοτήσεω ετησία των ελεκτικών φορέων. Η αρχή ελέγχου στέλνει μία γνωμοδότηση επί του ελέγχου στο τέλο του έτου κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου αναφέρει εκεί ποια είναι η άποψή τη σχετικά με το κατά πόσο τα συστήματα έχουν λειτουργήσει σωστά και αποτελεσματικά. Λοιπόν, αν έχουμε θετική τοποθέτηση του ελεκτικού φορέα που λέει ότι όλα τα συστήματα λειτουργούν σωστά, τότε μπορούμε να συναγάγουμε ότι μπορούμε να βασιστούμε στη διαδικασία πιστοποίησεω και ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας πολύ χαμηλός κίνδυνος ατασταλίας. Και η διαδικασία συνεχίζεται κατά τη διάρκεια όλης της περίοδου εφαρμογής μέχρι ότου λήξουν τα προγράμματα στο τέλος της περίοδου όπου υποβάλλονται τελικά λογιστικά στοιχεία, έχουμε τελική γνωμοδότηση ελεγκτική και πληρώνουμε τελικά ποσά οφείλονται. Αυτό είναι το παρόν σύστημα. Τώρα, ε, αν δούμε τι αναφέρεται στην πρόταση για την τροποποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού. Το βασικό άρθρο είναι το άρθρο 56. Εκεί υπάρχουν διάφορα σημαντικά στοιχεία. Υπάρχουν αντίκτυπο σε ό,τι αφορά τις απαιτήσει τροποποίησης του τρέχον συστήματος. Καταρχήν αναφέρεται ότι πρέπει να υπάρχει μία και μόνη διαχειριστική αρχή για οποιαδήποτε, για οποιαδήποτε ταμείο, για οποιαδήποτε πολιτική. Ο στόχος αυτής της α, ρύθμισης είναι ότι η λογοδοσία και η, η υπευθυνότητα θα πρέπει να, επομίζονται, να τις επομίζεται μόνο μια αρχή σε επίπεδο διαχείρισης. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία πιστοποίησης ώστε το κράτος μέλος να πιστοποιεί την ε, αρχή αυτή, δηλαδή να δείχνει την ικανοποίησή του για το ότι αυτή η αρχή έχει τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες για να μπορέσει να φέρει σε πέρας τον διαχειριστικό, του, διαχειριστικό ρόλο. Και η διαδικασία αυτή δεν θα πρέπει να είναι μία διαμιάς και μονάχα την πρώτη, στην αρχή της διαδικασίας διαδικασία, αλλά θα απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση, ώστε αν η διαχειριστική αρχή δεν εκπληρεί πλέον τα κριτήρια θα μπορούσε να, ε, να αποσυρθεί ή να ανασταλεί η πιστοποίηση. Τρίτο στοιχείο, να υπάρχει μια ετήσια δήλωση διαχειριστικού χαρακτήρα που υποβάλλεται από την ενιαία πιστοποιημένη αρχή κάθε χρόνο προς την Κομισιόν που θα συνδέεται με τους ετήσιους λογαριασμούς, ώστε ο ετήσιος η ετήσια δήλωση θα λέει ότι πράγματι οι ετήσιοι λογαριασμοί είναι αληθείς, αξιόπιστοι και ε, αντανακλούν την πραγματικότητα. Και έτσι θα φαίνεται ότι οι δαπάνες μέσα στους οι οποίες αναφέρονται στους λογαριασμούς αυτούς ήταν ε, νομότυπες και σωστές. Θα υπήρχε επίσης και μια ε, γνωμοδότηση λογιστικού ελέγχου σε σχέση με την ακρίβεια των λογαριασμών αλλά επίσης και σε σχέση με την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος και για την νομιμότητα και τακτικότητα των συναλλαγών αυτών που γίνονται. Και το τέταρτο καινοτόμο στοιχείο θα υπάρχει ετήσια εκαθάριση των λογαριασμών. Θα υποβάλλονται οι λογαριασμοί μαζί με την ετήσια διαχειριστική δήλωση και την ε, γνωμοδότηση λογιστικού ελέγχου και η Κομισιόν θα εξετάζει όλους αυτούς τους λογαριασμούς και θα παίρνει μια απόφαση για το αν αποδέχεται αυτούς τους λογαριασμούς, δηλαδή αν θεωρεί ότι αυτοί οι λογαριασμοί απεικονίζουν την πραγματικότητα και έχουν τη σωστή λογιστική απεικόνηση. Κάτι το οποίο περαιτέρω συνδέεται με τα έγγραφα αυτά τα οποία πρέπει να υποβληθούν θα είναι μια ετήσια σύνοψη των ελέγχων και λογιστικών ελέγχων που γίνονται κάθε χρόνο και αυτό θα είναι τμήμα του των εγγράφων που θα υποβάλλονται. Ποιες είναι τώρα οι αλλαγές οι οποίες απορρέουν από την εφαρμογή στις κατατομής ρυθμίσεις, στους κατατομής κανονισμούς σε σχέση με αυτό το οποίο παρουσίασα προηγουμένως ως το τρέχον σύστημα. Καταρχήν αντί να έχουμε τρεις αρχές, μία αρχή διαχείρισης, μία αρχή πιστοποίησης και μία αρχή ελέγχου, θα έχουμε δύο μοναχαρχές οι οποίες θα λαμβάνουν, θα έχουν κάποιο ρόλο. Θα έχουμε την αρχή διαχείρισης η οποία θα κάνει όλους τους ελέγχους πρώτου επίπεδου και στη συνέχεια θα λέει ποια είναι τα στοιχεία τα οποία πρέπει να τύχουν απόδοση εξόδων και θα έχουμε και την αρχή λογιστικού ελέγχου η οποία θα κάνει τα ίδια που κάνει τώρα, θα κάνει τον ex post έλεγχο και θα δίνει μια γνωμοδότηση περί λογιστικής ακρίβειας. Δεν έχουμε πλέον την πιστοποιητική αρχή επομένως στο ρόλο που έχει σήμερα. Δεύτερη αλλαγή είναι ότι θα περνούσαμε από το τωρινό σύστημα για την εκτίμηση της συμμόρφωσης σε ένα νέο σύστημα πιστοποίησης. Δεν είναι ριζικά διαφορετικό αυτό, αλλά θα έδινε την έμφαση στην πιστοποίηση μίας ενιαίας αρχής και όχι μίας εξέτασης του συνόλου του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου και έτσι θα υπάρχει μια συνεχής ευθύνη, δεν θα είναι μια μοναδική στιγμή που θα είναι υπεύθυνη αυτή η αρχή, θα πρέπει να υπάρχει μια πιστοποιούσα αρχή και μια πιστοποιούμενη αρχή. Η πιστοποιούσα αρχή θα παρακολουθεί την πιστοποιημένη αρχή σε όλη την διάρκεια της περίοδου προγραμματισμού. Τρίτη αλλαγή, η ετήσια δήλωση διαχείρισης, κάτι το οποίο δεν έχουμε αυτή τη στιγμή στους τωρινούς μας κανονισμούς, θα υπάρχει η πρόνοια μιας ε, ετήσιας διαχειριστικής δήλωσης που να συνοδεύει τους λογαριασμούς. Αντί να έχουμε λοιπόν πιστοποίηση των απαιτήσεων πληρωμών θα υπάρχει μια ετήσια δήλωση που θα λέει ότι όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στους ετήσιους λογαριασμούς ήταν ε, τυπικά σωστοί και επακριβείς. Και θα έχουμε στη συνέχεια τη διαδικασία του ε, τις ετήσιας εκαθάρισης λογαριασμών με την επίσημη απόφαση της Κομισιόν. Αν μπορέσω τώρα εν συντομία να σας πω τι θετικό θα προκύψει από αυτές τις αλλαγές. Αλλά σας πω και ποιοι είναι οι ελοχεύοντες κίνδυνοι για αυτές τις αλλαγές. Τα δυνητικά ωφέλη. Πρώτα απ' όλα θα υπάρξει μια εναρμόνιση σε μεγάλο βαθμό των προσεγγίσεων σε σχέση με την κοινή διαχείριση. Γιατί αυτό το σύστημα αν εφαρμοστεί στην πολιτική συνοχή θα είναι πολύ πιο κοντά στο σύστημα το οποίο εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή στο χώρο της αγροτικής πολιτικής για τον πρώτο πυλώνα εγγύσεων αλλά και για το δεύτερο πυλώνα αγροτικής ανάπτυξης. Αυτό λοιπόν θεωρείται ότι είναι ένα πλεονέκτημα το να έχουμε μια πιο ε, ομοιόμορφη διαδικασία για τα θέματα διαχειρισμέ... διαμοιρασμένης μάλλον διαχείρισης. Το να έχουμε μία και μόνη αρχή μπορεί να θεωρηθεί ότι εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει διάχυση ευθυνών. Εάν υπάρχει μόνο μία αρχή η οποία είναι υπεύθυνη και πρέπει να καταλήξει σε μία διοικητική και διαχειριστική δήλωση, είναι σαφές ότι εκεί βρίσκονται οι υπεύθυνοι και υπάρχει απόλυτη γραμμή λογοδοσίας. Υπάρχει επίσης πλεονέκτημα στο να έχουμε μια ετήσια διαχειριστική δήλωση, γιατί αυτό είναι το, το η συγκεκριμενοποίηση της ευθύνης. Ο διευθυντής της διαχειριστικής αρχής θα πρέπει πράγματι προσωπικά να υπογράψει το ότι έχουν γίνει οι κατάλληλοι και οι πρέποντες έλεγχοι και όλα τα ποσά έχουν ε, δαπανηθεί πρεπόντως είναι σαν τις ετήσιες εκθέσεις που υπογράφουν οι γενικοί διευθυντές στην Κομισιόν. Διατρέχεται λοιπόν από την ίδια αρχή ότι ο διαχειριστής θα πρέπει να έχει την ευθύνη του διαχειριζομένου και αυτό γίνεται με την υπογραφή μιας ετήσιας δήλωσης. Και μετά σε ό,τι αφορά την ετήσια διαδικασία εκαθάρισης, το πλεονέκτημα είναι ότι υπάρχει διαφάνεια. Γιατί κλείνουν οι λογαριασμοί κάθε χρόνο, αντί να κλείνουν τώρα όπως τώρα. Μόνο στο τέλος της προγραμματικής περίοδου, εννέα χρόνια μετά από την αρχή. Κλείνοντας τους λογαριασμούς κάθε χρόνο, έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και μπορείτε να δείτε τι δαπανήθηκε πιο χρόνο και για ποια ενέργεια. Επίσης, ανοίγει το δρόμο στο να έχουμε μια συντομότερη περίοδο για την οποία οι τελικοί αποδέκτες θα πρέπει να κρατάνε τα παραστατικά και δικαιολογητικά έγγραφα. Αυτό δεν λέγεται στην πρόταση για το δημοσιονομικό κανονισμό, αλλά είναι δυνητική απόρρια αυτού του κανονισμού που θα κάνει πιο εύκολο να έχουμε κανόνες σε τομεακό επίπεδο που θα μειώνουν τον χρόνο για τον οποίο θα πρέπει να κρατάνε τα παραστατικά για επιθεώρηση οι τελικοί αποδέκτες. Αυτά λοιπόν τα θετικά στοιχεία που βλέπουμε για την βελτίωση της διαδικασίας ελέγχου και εξασφάλισης της διαδικασίας. Από την κινδυνική πλευρά, κάτι το οποίο προέκυψε από τις συζητήσεις με τα κάτι μέλη, είναι ότι η αλλαγή από ένα σύστημα το οποίο γνωρίζουν σε ένα σύστημα το οποίο δεν γνωρίζουν, αυτό ήδη περιέχει κάποιους κινδύνους. Είπαν τα κράτη-μέλη τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει μια μεγάλη επένδυση για να μπορέσουν να υλοποιήσουν ένα σύστημα το οποίο θα συμμορφώνεται με τις διατάξεις οι οποίες είχαν τεθεί για την περίοδο 2007 μέχρι 2013 χρειάστηκε να κάνουμε μια πάρα πολύ δύσκολη και επαχθή και πολυδάπανη διαδικασία συμμόρφωσης με ελέγχους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τροποποίηση επί τη βάση των προτάσεων και των συστάσεων της Κομισιόν και έχουμε τώρα συστήματα τα οποία λειτουργούν μια χαρά. Και εκεί που λειτουργούν μια χαρά τα συστήματα, εάν τα αλλάξουν, αν αλλάξει η αρχιτεκτονική ελέγχου, ανησυχούν γιατί θα πρέπει να περάσουμε μια διαδικασία προσαρμογών και αλλαγών, να χρησιμοποιήσουν νέους φορείς οι οποίοι θα εμπλέκονται, να έχουν νέα εγχειρίδια, να επανεκπαιδεύσουν το προσωπικό τους κτλ. Όλα αυτά είναι ένας κίνδυνος μόνο και μόνο γιατί πρέπει να αλλάξουμε από μία αρχιτεκτονική ελέγχου σε μία άλλη αρχιτεκτονική ελέγχου. Ο δεύτερος τομέας όπου θα έλεγα ότι υπάρχει σημαντική ανησυχία κινδύνου είναι για το διοικητικό άχθος. Θεωρούν ότι μπορεί να προκύψει αυξημένο διοικητικό άχθος λόγω του ότι οι παραδοσιακοί θα πρέπει να κάνουν ετήσιους λογαριασμούς, θα πρέπει να παρουσιάσουν μια αιτήσια διαχειριστική δήλωση, όλα αυτά είναι νέα στοιχεία και θεωρούν ότι θα είναι προβληματικά ενδεχομένω τα στοιχεία αυτά και επίσης γιατί θα υπάρχει αυτός ο συνεχής ρόλος της πιστοποιούσας αρχής που φαίνεται να είναι μία ακόμα πρόσθετη στρώση στο σύστημα. Αυτά λοιπόν τα διάφορα στοιχεία τα οποία αναφέρθηκαν, τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν και να τα ζυγίσουμε τα υπέρ και τα κατά του συστήματος σε ένα σεμινάριο το οποίο οργανώθηκε από την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακών Θεμάτων μαζί με τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμών και τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης είχαμε την ευκαιρία να προβούμε σε μια ανταλλαγή απόψε με τα κράτη-μέλη για τα θέματα αυτά. Και αυτά ήταν κάποια θέματα τα οποία προέκυψαν από αυτό το σεμινάριο. Από την πλευρά της Κομισιόν. Ενώ μπορούμε να δούμε ότι στις διαδικασίες αυτές της συζήτησης μπορεί να υπάρχει ανάγκη να κάνουμε κάποιες προσαρμογές, θεωρούμε ότι είναι κομβικά ορισμένα στοιχεία που αφορούν την ενίσχυση του συστήματος. Το να έχουμε καταρχήν μια αιτήσια δήλωση διοικητικής διαχείρισης, να έχουμε διαφορετικές διαδικασίες που να οδηγούν σε ένα έγγραφο μονάχα σε αιτήσιο επίπεδο που να το υπογράφει ο επικεφαλής της διαχειριστικής αρχής, αυτό θα ενισχύσει το σύστημα. Δεύτερον, βλέπουμε να υπάρχει ένα πλεονέκτημα αν υπάρχει ο συνεχιζόμενος ρόλος μιας πιστοποιούσας αρχής, όχι μονάχα να ελέγχει τη συμμόρφωση στην αρχή, αλλά το να υπευθυνοποιούνται τα κράτη-μέλη για την εποπτεία και την επιθεώρηση του έργου της διοικητικής αρχής, ώστε εάν δεν έχει πλέον τις απαραίτητες ικανότητες η αρχή αυτή, θα πρέπει να αποσύρουν την πιστοποίησή της. Τρίτον και πλέον σημαντικών, βλέπουμε ένα πλεονέκτημα στην εξασφάλιση του ότι οι διαβεβαιώσεις που παίρνουμε από τα κρατη μέσω των ελεγκτικών τους αρχών ότι αυτές οι διαβεβαιώσεις αφορούν ακριβώς τις ε, δαπάνες που οδηγούν σε πληρωμές από την Κομισιόν. Όταν λέει η Εθνική Αρχή ότι τα έλεγξα αυτά και είμαι ικανοποιημένο ότι ήταν νομότυπα και επακριβή όλα αυτά τα στοιχεία, τότε ξέρουμε και εμείς ότι οι δικές μας πληρωμές είναι εξασφαλισμένες. Όταν λοιπόν εμείς έχουμε να κοιτάξουμε τις ε, πληρωμές που κάνουμε σε ένα οικονομικό έτος, θα πρέπει να έχουμε έναν τρόπο να τις συνδέσουμε σε ένα, με ένα οικονομικό έτος στο κράτος μέλος, το οποίο αντιστοιχεί ακριβώς σε αυτή τη χρονική περίοδο και αυτό είναι πιο καλό και για μας και βοηθάει περισσότερο τη διαδικασία απαλλαγής να έχουμε αυτή την ε, σύνδεση εξασφαλίσεων από το κράτος μέλος στην Κομισιόν που θα ενισχύσει το σύστημα. Λέω να σταματήσω εδώ κυρία Πρόεδρε. Αλλά φυσικά μπορώ να σας δώσω και λεπτομέρειες περαιτέρω εάν το επιθυμείτε. Ευχαριστώ να ενημερώσω τον συνάδελφο ότι ο κ. Μάρτιν είναι ε, ο ότι υποδιευθυντής ε, σε ό,τι αφορά την πολιτική συνοχή στη διεύθυνση επικοινωνίας. Και τώρα να δώσω τον λόγο στον εισηγητή μας, τον Γιάνν Όλμπριχτ, να μας κάνει και αυτό στη δική του παρουσίαση, να ακούσουμε τα σχόλιά του. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, όντως, ο γενικός ε, κανονισμός είναι κάτι το οποίο δεν συζητάμε σε πρώτη φάση στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, γιατί φαίνεται ότι δεν έχει περιφερειακή διάσταση, μόνο διάσταση από πλευράς προπολογισμού. Να πω, και το λέω αυτό μάλλον με την εξαιτή μου εμπειρία, κατά δεύτερον ότι είναι πάρα πολύ περίπλοκο το πρόβλημα. Γιατί εξ αρχής συζητιόταν το κατά πόσον ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ως θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να επένδουμε σε κάποια άρθρα ή να δώσουμε τη δυνατότητα να ανοίξουν όλα τα άρθρα. Το κείμενο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που προτάθηκε μάλλον τον ε, Δεκέμβριο του 2010, αποτελεί την πρόταση βάσει της οποίας αποφασίζει και προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μάλλον πρόκειται για, συ, για συναπόφαση. Το, τμήμα της, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το προετοιμάζουν η Επιτροπή Προπολογισμών και Ελέγχου Προπολογισμού. Γι' αυτό λοιπόν τώρα θα πρέπει να συνενώσουμε τα έγγραφα εργασίας που έχουν προετοιμάσει και η κυρία Γκρέσλε και τον κύριο Δεβελίνη που πλευρά τη Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού. Άρα λοιπόν σήμερα έχουμε καταρχά τι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά δεύτερον την αντίδραση του Κοινοβουλίου και κατά τρίτον γνωρίζουμε ότι αυτή είναι η στάση των κρατών μελών. Άρα και τα τρία αυτά στοιχεία μας φέρνουν σε μια πολύ δύσκολη θέση, γιατί είναι δύσκολο να βρούμε συμφωνία και κοινό τόπο. Ο βασικός δημοσιονομικός κανονισμός δεν αφορά μόνο την περιφερειακή πολιτική. Αφορά όλο το οικονομικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τμήμα αυτού είναι η κοινή διαχείριση. στην ε, έμεση διαχείριση του κανονισμού. Ο απότερος στόχος, η γενική ιδέα εξ αρχής ήταν, από ήταν να απλοποιήσουμε το σύστημα, το οποίο πολύ συχνά καταλήγει να περιπλέκει παραπάνω το σύστημα, αλλά εν πάση περιπτώσει σκοπός μας ήταν να απλοποιήσουμε το σύστημα. Είναι σημαντικό όμως επίσης να διευκρινιστεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο όλο σύστημα. Άρα στον κανονισμό βλέπουμε την πρόταση απλοποίησης του, της διασφάλισης του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του ορισμού του ρόλου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών. Αυτή ήταν η βασική ιδέα. Αυτό θέλαμε μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας, να διευκρινιστεί ο ρόλος όλων των θεσμικών οργάνων. Στο κείμενο τώρα πλέον τι βρίσκουμε. Προτάσεις να αλλάξουν περίπου 200 άρθρα. Αυτή είναι η πρόταση τώρα. Σε ό,τι αφορά τα προβλήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και του αποδεκτού επίπεδου κινδύνου. Μάλλον του περιθωρίου σφάλματος. Μπορούμε να το συζητήσουμε στο Κοινοβούλιο. Τι σημαίνει αυτό για τους μακροοικονομολόγους. Τι εννοούμε από δεκτό περιθώριο ασφαλμάτων. Και δεν είμαι εγώ οικονομολόγος, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι ούτε οι οικονομολόγοι συμφωνούν μεταξύ τους. Και ασφαλώς και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η δυνατότητα ε, ευελιξίας από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα όρια της ευελιξίας αυτής και ασφαλώς το θέμα και το πρόβλημα των, ε, της έμεσης και άμεσης διαχείρισης, γιατί εμείς σήμερα συζητάμε την έμεση διαχείριση. Αυτό που μόλις μας περιέγραψαν και κάποιοι συνάδελφοι από την Επιτροπή Προπολογισμών και Ελέγχου του Προπολογισμού συμφωνούν σε πολλές περιπτώσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα θα μπούμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση γιατί εν γέννη η Επιτροπή Προϋπολογισμού, οι εισηγητές δηλαδή, θέλουν να ενισχύσουν σε πρώτη φάση το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά δεύτερον, και από τις δύο επιτροπές οι εισηγητές θέλουν να διευκρινιστεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να μην έχει πάρα πολλές δυνατότητες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι περιορισμένο, περιορισμένος ο ρόλος της και να οριστεί η έμεση διαχείριση, για παράδειγμα το EIB και το χρηματοπιστωτικά μέσα. Σε ό,τι αφορά... Σε ό,τι αφορά την κοινή διαχείριση. Δύο θέματα. Σε ό,τι αφορά και τη σύγκριση με τα σημερινά συστήματα. Η, η μεγάλη πρόκληση είναι η εξή. Αυτό που παρατηρούμε σήμερα είναι το εξή. Η αποδοτικότητα του συστήματος βελτιώνεται διαρκώς. Εφόσον λοιπόν βελτιώνεται, θα έπρεπε να το αλλάξουμε. Αυτό συχνά μας λένε τα κράτη-μέλη. Αν το σύστημα τα πηγαίνει καλά και περιορίζεται το περιόριο σφάλματος, πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα και σε ποιο βαθμό. Και πώς ε, θα αποφύγουμε υπερβολικές περιπλοκές. Χωρίς να χάσουμε τα θετικά αποτελέσματα τα οποία που έχουμε πετύχει. Γιατί αυτό που βλέπουμε στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού είναι ότι υπάρχουν πολύ καλά, σαφή, καλά θετικά αποτελέσματα. Γιατί αλλάζουμε λοιπόν το σύστημα. Η πρώτη ερώτηση είναι γιατί να το αλλάξουμε. Και επίση, ποιε είναι οι αλλαγέ οι οποίε είναι αναπόφευκτε, απόλυτα απαραίτητε. Έχω την εντύπωση ότι κινούμαστε προ την πλευρά τη πολιτική απόφαση. τι θα πρέπει να αλλάξει απαραίτητος και τι δεν χρειάζεται απαραίτητα να αλλάξει. Η δεύτερη ιδέα πίσω από αυτό. Ότι ίσως θα έπρεπε να κοιτάξουμε λίγο τις εμπειρίες μας από το CAP και να τις εφαρμόσουμε. Είναι διαφορετικό το CAP. Κάποια α, από την εμπειρία μας από τη μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής. Ακόμα και στην ομάδα μας, ακόμα και σήμερα, ο εισηγητή ε, για την απαλλαγή συμφώνησε μόλις να αλλάξει την έκφραση που αναφέρει ότι η εναρμόνιση της κοινή αγροτικής πολιτικής και να την κάνει, μάλλον να αλλάξει την διατύπωση και να την ε, κάνει να αναφέρει διευκρίνηση μεταξύ κοινή γεωργικής πολιτική. Πρέπει να δούμε λοιπόν ποιες κοινέ εμπειρίε υπάρχουν για τις δύο αυτές πολιτικές. Καταρχάς το πρόβλημα της ε, δομής και της οργάνωσης και ότι θα πρέπει να υπάρχει μικρότερος αριθμός θεσμικών οργάνων. Το πρώτο, η πρώτη αρχή πιστοποίησης, οι συγκητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχαν προτείνει να είναι υπεύθυνη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πιστοποίηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τα κράτη-μέλη να έχουν μία αρχή πιστοποίησης η οποία θα είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τη λειτουργία των ε, πιστοποιημένων σωμάτων. Τα πιστοποιημένα σώματα τα οποία θα αντικαταστήσουν τις υπηρεσίες διαχείρισης όπως μας εξήγησε και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, θα πιστοποιούνται λοιπόν και θα ελέγχονται κατά τη διάρκεια της περίοδου από ε, μια κεντρική υπηρεσία. Τι γίνεται σε ό,τι αφορά την πιστοποίηση στην κοινή γεωργική πολιτική. Αυτό αποτελεί μια ομοιότητα. Το πρόβλημα της ε, πιστοποίησης και των πιστοποιημένων υπηρεσιών. Να σας υπενθυμίσω ότι συνεχίζεται η συζήτηση στην Επιτροπή Ελέγχου του Προεπλογισμού σε ό,τι αφορά την Εθνική Δήλωση Ασφάλειας. Και την ευχή του Ευρωκοινοβουλίου να εγκριθεί από τα κράτη-μέλη, η οποία ασφαλώς και είναι φρούδα. Αυτό που παρατηρούμε λοιπόν σήμερα είναι το εξή. Ότι τα πιστοποιημένα σώματα θα είναι υπεύθυνα για την δήλωση διαχείρισης. Αυτή θα είναι υπεύθυνη. Και φυσικά η γενικότερη τάση που παρατηρούμε σήμερα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει, προτείνει να δώσει πιο πολλές αρμοδιότητες στα κράτη-μέλη ασφαλώς. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να πιστοποιούν τις υπηρεσίες και μέσω των πιστοποιημένων υπηρεσιών θα πρέπει να ελέγχουν του πιστοποιημένου τα κράτη-μέλη και πάλι. Είναι αρμοδιότητα του, κρατου, του μέλου. Μία δεύτερη μεγάλη αλλαγή. Και αυτό είναι πρόβλημα του εθνικού λογιστικού έτου. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα, γιατί ποια είναι η προθεσμία κατά την οποία θα ανασταλούν οι πληρωμές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να είναι η 30 Σεπτεμβρίου η ημερομηνία αυτή. Το λογιστικό έτος δηλαδή να ξεκινάει από τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους. Αλλά το λογιστικό έτος είναι από τον Ιανουάριο προς το, το έτος στον προϋπολογισμό, στον προϋπολογισμό, στο δημοσιονομικό έτος, είναι από Ιανουάριο μέχρι Δεκέμβριο. Για παράδειγμα, το 2011 οι πληρωμές αναστέλλονται τέλος ε, Σεπτεμβρίου και μετά θα έχουμε αξιώσεις για πληρωμές οι οποίες θα περάσουν στο επόμενο έτος γιατί θα εξεταστούν στο επόμενο δημοσιονομικό έτος. Άρα ερωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το συζητήσαμε αυτό και σήμερα. Από πού έρχεται αυτό το σύστημα και πάλι από την ΚΑΠ. Γιατί αυτό το σύστημα από Σεπτέμβριο σε Σεπτέμβριο λειτουργεί στην ΚΑΠ. Άρα η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για καλύτερο έλεγχο Ίσως θα μπορούσε να μας εξηγήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μήπως κάτι κατάλαβα λάθος είναι ότι αν τελειώσουν οι πληρωμές στα τέλη του Σεπτεμβρίου αυτό τι σημαίνει ότι η ετήσια έκθεση θα βασίζεται στις πληροφορίες για τις πληρωμές 9 μηνών του δημοσιονομικού έτους. Άρα θα δοθούν οι πληροφορίες για την ποιότητα των πληρωμών μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου. Άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει τις πληροφορίες από την δήλωση διαχείριση στα τέλη του χρόνου. Δηλαδή τρει μήνε αργότερα, με τρει μήνε καθυστέρηση. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει τι πληροφορίε για την ετήσια έκθεση ένα χρόνο αργότερα. Αυτή είναι λοιπόν μια βασική αλλαγή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προτείνει να περιοριστεί ο χρόνος για την κατάθεση της έκθεσης. Να λαμβάνει τι πληροφορίε αυτές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε λιγότερο χρονικό διάστημα με ε, διαφορετικό επίπεδο ελέγχου όμω. Αλλά πιο γρήγορα να έχει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις πληροφορίες αυτές τις απαραίτητες στα τέλη του χρόνου. Θα αλλάξει αυτό το σύστημα χορήγησης απαλλαγής. Όχι ιδιαίτερα. Θα αλλάξει την ποιότητα της απαλλαγής, όχι την ημερομηνία της απαλλαγής. Γιατί αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στα τέλη του δημοσιονομικού έτους, το Δεκέμβριο δηλαδή, τις απαραίτητες πληροφορίες βάσει Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προετοιμάσει τα έγγραφά της θα διαβιβάσει τις πληροφορίες στο ελεκτικό συνέδριο και άρα τους επόμενους μήνες του επόμενου έτους θα ξεκινήσει στα τέλη του επόμενου έτους του δημοσιονομικού έτους θα ξεκινήσει η διαδικασία χορήγησης απαλλαγής. Άρα τι προτείνουμε, να έχουμε το λογιστικό έτος το οποίο θα λέγει τέλη Σεπτεμβρίου, να έχουμε το δημοσιονομικό έτος το οποίο θα είναι το έτος για την χορήγηση της απαλλαγής. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία. Καταρχάς λοιπόν η πρόταση απλοποίηση στο σύστημα για το ρόλο των θεσμικών οργάνων και να υπάρχει μία αρχή πιστοποίηση στα κράτη-μέλη που θα είναι υπεύθυνη για την πιστοποίηση και την εποπτεία των πιστοποιούμενων υπηρεσιών και τα πιστοποιούμενα αυτά τμήματα, σώματα θα κάνουν την σχετική δήλωση διαχείρισης και θα πιστοποιείται αυτή από τις αρμόδιες αρχές και κατά δεύτερον Δεύτερο στοιχείο, ότι το λογιστικό έτος φυσικά θα έχουμε διάφορο, διαφορετικούς τρόπους ελέγχου της ποιότητας των δαπανών. Αυτό είναι τμήμα της κοινή διαχείρισης. Άρα υπάρχει μια σαφής ε, πρόταση να ασπαστούμε κάποια ε, προγράμματα από την ΚΑΠ, χωρίς όμως τον πολιτική χαρακτήρα. Ευχαριστούμε, Γιάν. Έχουμε σκυρώδεις συγγητές που θέλουν να πάρουν το λόγο. Και Γκάι δεν είναι εδώ. Ρίκα Μάνα, θες να πεις κάτι. Φρανσουά Αλφονζή, θες να πεις κάτι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχουμε τρεις στόχους. Πρώτος, η καλύτερη απλοποίηση είναι η συνέχεια. Είναι ουσιαστικό αυτό. Αν ακολουθήσουμε πολύ τεχνοκρατική προσέγγιση, καμιά φορά δεν το διακρίνουμε αυτό. Δεύτερον, αποτεσματικότητα των μέσων, φαινόμενο μόχλευση. Χρειάζεται θέτηση κανονισμού. Για να υπάρχουν, ε, ε, να έχουμε το φαινόμενο μόχλευση τη Ευρωπαϊκή Τάξη Επενδύσεων κλπ. και τη μελλοντική πολιτική τη Ευρώπη, χρειάζεται ο δέον ε, κανονισμό. Και τέλο, είναι αναγκαίο. Όλοι το ζητούν ομόφωνα, όσοι έχουν με σχέση με την ευρωπαϊκή διοίκηση θέλουν απλούστευση και αναλογικότητα των διαδικασιών. Εν συγκρίση με τα διακυβευόμενα του κάθε τομέα. Θα έπρεπε να υπάρχει ενιαίο κανόνα είτε δίνουν χίλια, είτε χιλιάδε ε, ευρώ, δεν ξέρω. Χρειάζεται αναλογικότητα. Προανέφερα τρει άξονε. Πράγματι χρειάζεται ένα κανονισμό που συμπεριλαμβάνει αυτό το φαινόμενο μόχλευσης σε όλες τις δυνατότητες υποστήριξης και στα πλαίσια εταιρικών σχέσεων. Να υπάρχει σωστή συνεργασία επί τόπου. Όμως προσοχή, όταν τροποποιείται ένας κανονισμός, ξεκινά μια νέα περιπέτεια για τους δικαιούχους. Πρέπει να ενημερωθούν, ούτως ώστε να μπορέσουν να αντιληφθούν όλες τις μικρολεπτομέρειες και συνεχεία το προσωπικό να είναι καταρτισμένο για να ετοιμάζει τα έγγραφα σε κατάσταση τέτοια που είναι αποδεκτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, στη μεταρρύθμιση, αλλά προσοχή σε πολλέ μεταρρυθμίσει που θα μπορούσαν να σκοτώσουν την μεταρρύθμιση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μάρκο Πίμπελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω ένα ερώτημα προς την Κομισιόν, αλλά και για τον Γιάνν Όλμπριχτ επίσης. Εγώ θεωρούσα ότι σε κάποια κράτη-μέλη είχαμε προβλήματα μονάχα και εκεί θα υπήρχε κάποια ανάγκη βελτίωση του, στοιχείου, του συστήματος και είχα πάντα την ε, προσδοκία από την Κομισιόν ότι για τα θέματα πιστοποίησης θα μπορούσε η ίδια να είναι πιο υπεύθυνη και να αναλάβανε την ευθύνη της πιστοποίησης. Εγώ φυσικά θα βλέπω τα πράγματα να είναι πιο θετικά όταν υπάρχει μία ενία αρχή που να αναλαμβάνει την ευθύνη. Αυτό το κάνει το σύστημα πιο αποδοτικό, αλλά ανησυχώ ήδη γιατί όταν ένα κράτος μέλος το οποίο έχει δείξει στο παρελθόν ότι τα στοιχεία του δεν είναι επακριβή, αν δώσουμε σε αυτό το κράτος την απόλυτη εμπιστοσύνη ώστε μόνο του να πιστοποιήσει τις δικές του εποπτικές αρχές, αυτό με ανησυχεί. Θα ήθελα να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ανεξαρτησία και πολύ πιο έντονη συμμετοχή της Κομισιόν στη διαδικασία πιστοποίησης και θα ήθελα επίσης να υπάρχει μια διαδικασία που εξασφαλίζει ότι αν έχει πιστοποιηθεί μία αρχή θα έχει μια μεγαλύτερη ε, μεν ε, μια μεγαλύτερη ελευθερία να μην υποβάλει τόσε πολλέ εκθέσει ώστε να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε την προσοχή μα αποκλειστικά και μόνο στα μαύρα πρόβατα, εκεί που θεωρούμε ότι υπάρχουν προβλήματα. Δεν βλέπω λοιπόν να γίνεται αυτό με ένα σύστημα το οποίο, από το οποίο αφαιρείται η, η υπευθυνότητα τη Ευρωπαϊκή πλευρά και επαφίονται τα πάντα στα κράτη-μέλη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω θα, θα ξεκινήσει μεγάλη συζήτηση και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Ελίζαπεθ Σρέντερ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Και εγώ προσπάθησα να καταλάβω όλα αυτά τα οποία ανέφερε η Κομισιόν, αλλά βρίσκω πολύ σημαντικά αυτά που ανέφερε ο Γιάννη. Εγώ έχω τώρα πολλά ερωτήματα να σας θέσω. Εγώ συμμερίζομαι αυτά που είπε ο Μάρκους Πίπερ, ότι η Κομισιόν αυτή τη στιγμή χάνει την ευθύνη που είχε για το σύστημα και ερχόμαστε και στο ερώτημα αυτό του Γιάννη. Τότε, όταν η δική μας Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ρωτάει την Κομισιόν να πει πόσα είναι τα πόσο τμήμα του προπολογισμού δεν εκτελέστηκε σωστά, τι θα μας πει η Κομισιόν. Δεν έχουμε ιδέα. Μόνο τα κράτη-μέλη το ξέρουν αυτό. Δηλαδή, μπορούμε να φανταστούμε μια τέτοια κατάσταση. Τι θα κάνουμε τότε. Και επίσης, σε όλο αυτό το σύστημα από τη δική μου πλευρά, ή τουλάχιστον δεν το έχω καταλάβει ακόμα, δεν υπάρχει κάποιο σύστημα ελέγχου της Κομισιόν. Πώς μπορούμε εμείς λοιπόν να ασκήσουμε έλεγχο σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Κομισιόν για το ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια έχουν πάει εκεί που έπρεπε να πάνε. Και είναι λεφτά του Ευρωπαίου φορολογούμενου. Είναι πολύ δύσκολο από τη μια πλευρά να έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία και από την άλλη πλευρά να έχουμε μεγαλύτερη ευθύνη. Εγώ έχω την εντύπωση ότι η Κομισιόν τραβάει την ουρά της λιγάκι από το σύστημα. Πρέπει λοιπόν να δούμε αν θα υπάρξουν συνέπειες από αυτό. Αλλά η Κομισιόν μου φαίνεται ότι δεν θα έχει τη δυνατότητα να κάνει κανένα έλεγχο. Έχει μόνο τη δυνατότητα να κάνει ελέγχους ad hoc και τίποτα παραπάνω. Φαντάζομαι ότι στο σύστημα θα προβλέπετε ότι οι αρμόδιες αρχές, εάν προσκληθούν από την Κομισιόν, θα έχουν πάντα τα έγγραφα και τα παραστατικά τα οποία απαιτούνται για να υπάρξει έλεγχος. Δεύτερον, υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία κάπως αποκρύπτονται μέσα σε ένα τέτοιο σύστημα. Το ερώτημα του τι γίνεται με τις περιφέρειες στο σύστημα αυτό. Η ισχυρή αυτή εξουσία της ε, αρχής της διαχειριστικής σημαίνει σε τελική ανάλυση μια ισχυρή κεντροποίηση του συστήματος και το άλλο ερώτημα το οποίο ανέφερε ο κύριος Όλμπρεχτ. Τι θα κάνουμε τώρα με τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα προκύψουν στο μέλλον αν θέλουμε να έχουμε μια τόσο πλήρη έκθεση για όλα αυτά τα θέματα. Υπάρχουν και χρηματοδοτήσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το σύστημα. πώ θα αντιμετωπιστούν αυτέ από ελεγκτική πλευρά. Και το τελευταίο ερώτημα, τι θα το κάνετε αυτό για προγράμματα τα οποία είναι διαμεθοριακού χαρακτήρα. Όταν έχετε ένα σύστημα το οποίο είναι τόσο στενά εθνικό, τι θα γίνει με διαμεθοριακού χαρακτήρα προγράμματα, με κοινά ευρωπαϊκά προγράμματα που χρειάζεται να υπάρχουν κοινέ ευρωπαϊκέ αρχέ. Υπάρχει μια πρόσθετη διαδικασία. Πώ θα λειτουργήσει λοιπόν αυτό το πράγμα. Έχουμε προγράμματα στα διαρθρωτικά ταμεία τα οποία είναι καθαρά εθνικού χαρακτήρα και έχουμε και διαμεθοριακά προγράμματα. Τι θα γίνει σε αυτήν την περίπτωση, ποιο θα τα ελέγχει αυτά τα προγράμματα. Αυτά είναι λοιπόν ερωτήματα τα οποία εγώ θέλω να θέσω και θα ήθελα να έχω μια απάντηση γιατί δεν βλέπω πώς θα λειτουργήσει σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν είμαι απόλυτα πεπισμένη λοιπόν ότι θα μπορέσουν όλα αυτά να λειτουργήσουν σωστά. Κατανοώ την πρόθεση της απλοποίησης αλλά υπάρχουν αυτά τα οποία είπε ο Μάρκους Πίπερ, ότι με τον τρόπο αυτό η, η Κομισιόν κάνει πάσα τα προβλήματα στα κράτη-μέλη και επομένως θα χρειάζεται να ελέγχουμε 27 κράτη-μέλη χωριστά για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται με τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ο Βανίστερο έχει το λόγο. Eh, Όντως, ε, στην κλίμακα, στις κλίμακες που ξέρουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις αυτόνομες περιφέρειες, στην περιφερειακή, τοπικό επίπεδο, στα εθνικά κρατημέλη. Όντως θα πρέπει να υπάρχει σε αυτά τα επίπεδα καλή κατανομή των ε, αρμοδιοτήτων. Και εγώ έχω αμφιβολίες και σε ό,τι αφορά να, να ανατεθεί η διαδικασία πιστοποίηση στα κρατημέλη. μελη γιατί είναι μια διαδικασία εκμάθησης Εγώ θα ήμουν υπέρ του να γίνεται αυτή η διαδικασία πιστοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αν υπάρχουν προβλήματα, να μην πιστοποιούνται οι οργανώσει να ακολουθήσουμε μια γραμμή ποιότητας και να μην έχουμε τις ε, απίθανες συζητήσει που γίνονται και τώρα στην, ε, στον έλεγχο των προπολογισμού. Κατά δεύτερον, σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση, αυτό γίνεται σε εθνικό επίπεδο και εγώ είμαι υπέρ της εθνικής ε, δήλωσης. Εγώ θεωρώ ότι θα ενισχύσει, το, θα μας βοηθήσει. Τώρα για την, τα προγράμματα ευρωπαϊκής διαχείρισης και σε ό,τι αφορά και την κοινή διαχείριση. Να μην τα μπλέκουμε αυτά. Γιατί αυτό θα ήταν μεγάλο σφάλμα. Το shared management είναι πάρα πολύ ιδιότυπο σύστημα. Και έτσι θα πρέπει να μεταφράζεται για τη διαδικασία τώρα. Είναι λίγο περίεργο. Κάνουμε αυτή τη συζήτηση για τον δημοσιονομικό κανονισμό ενώ μας ε, αφορά τόσο έντονα, αφορά τους κανονισμούς μας, τον... γιατί δεν έχουμε το περάρθρο 50. Γιατί δεν έχουμε αρμοδιότητα στην Επιτροπή, γιατί δεν έχουμε τέτοιες αρμοδιότητες. Έχω την εντύπωση ότι κάποια πράγματα μπορούν να πάνε τελείως λάθος. Τη στιγμή που δεν μπορεί κανείς ε, να επηρεάσει την κατάσταση. Έχουμε μία γνώμη απλά. Ίσως θα μπορούσε να μας σχολιάσει η πρόεδρος το πώς θα συνεχιστεί η διαδικασία τους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ, Λαμπέρ. Άλλος της, αγορεύει, βούλετε. μία, έχω τρία ερωτήματα, απευθύνοντας αυτά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς τον Γιάννη. Σύντομο σχόλιο. Στην περίπτωση που έθεσε η Ελίζα Στρέντερ τη ε, εδαφική συνεργασία, πώ θα λειτουργήσει το σύστημα. Δεύτερο ερώτημα. Για το δινηρό και χρονοβόρο θέμα τη αξιολογήσεω συμμόρφωση ε, που εσεί και ο Νίκολα ήταν υπεύθυνοι γι' αυτό για την περίοδο 2007-2013. Σε τι βαθμό μπορεί να ισχύει αυτή η αξιολόγηση και στο μέλλον με όλε τι αλλαγέ. Τρίτο ερώτημα μήπως καταλάβω αυτό που παρουσιάζετε. Πότε θα έρθει η στιγμή κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει κατά πόσο λειτουργεί σωστά το σύστημα ελέγχου και εποπτείας των κρατών μελών και κατά πόσο η αναδιάθρωσή του έχει γίνει με το σωστό τρόπο. Ο Νίκολας πρώτος ή εσύ πρώτος Γιάννη. Ο Γιάννη, να πάρω το λόγο τώρα για να ακούσω και την απάντηση στον όσο θα πω τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνοντα υπόψη τα σχόλιά σου. Και εγώ την ίδια εντύπωση σχημάτισα στην αρχή, ότι η εκχώρηση ευθυνών αφορούσε μόνο τα κράτη-μέλη. Όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να τα εξετάζουμε από κοινού, ταυτόχρονα. Αν θέλουμε να πλουστεύσουμε την κατάσταση και να μειώσουμε τον αριθμό των θεσμικών φορέων, Ποιο είναι το πρόβλημα για αυτή η περίπτωση. Ποιο σύστημα πιστοποίησης υπάρχει για κάτι που είναι απλουστευμένο. Δηλαδή υπάρχει συνάρτηση του αριθμού των θεσμικών φορέων με την διαπίστευση. Θέλουμε απλούστευση. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Εντάξει. Για τα κράτη-μέλη τώρα. Ο πιστοποιημένο φορέας θα είναι σε εθνικό επίπεδο, περιφερειακό επίπεδο. Αυτό εξαρτάται το κράτο μέλο θα αποφασίσει το κάτω μέλος και σύμφωνα με το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το θέμα είναι το εξή. Αν έχουμε πιστοποιημένους φορείς που είναι επίφθηνοι για επιχειρησιακά προγράμματα, ποιος κάνει την πιστοποίηση. Και όχι μόνο αυτό. Διότι διαπίστευση, πιστοποίηση τι σημαίνει. Ότι αυτό δεν είναι μόνο μία απόφαση, αλλά είναι αποτέλεσμα συνεχούς ελέγχου. Χρειάζεται η διοίκηση να παρακολουθεί συνεχώς κάθε πιστοποιημένο τομέα ε, φορέας σε κάθε κράτος Στις Βρυξέλλες θα υπάρχει ειδικό τμήμα που συνεχώς θα παρακολουθεί 200 πιστοποιημένους φορείς. Νομίζω ότι θα έχουμε περίπλοκη απλούστευση εν τη αυτή περίπτωση. Το θέμα είναι το εξής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αποσυρθεί από το πεδίο της μάχης. Εδώ είναι και το ερώτημα της Πρόεδρου. Πότε ελέγχει και διαπιστώνει τα πράγματα πηγαίνουν καλά είτε όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουν πρώτα πιστοποίηση. Ευθύνη των κρατών μελών. Επόμενο στάδιο. Όλες τις πληρωμές για τη λειτουργία του συστήματος και τη δήλωση της διαχείρισης. Ο πιστοποιημένος φορέας Λέει, μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι τα πάντα είναι καλά. Και αυτό είναι η αρχή, δεν το τέλος. Μετά, πάει αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πάει σαφής δήλωση ότι εγώ είμαι υπεύθυνο. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίρνει αυτό το έγγραφο και αν κάτι δεν πάει καλά, είναι σαφές ποιος είναι υπεύθυνο. Διότι κάποιο υπέγραψε ότι τα πάντα είναι μια χαρά. Στην αρχή αυτό περιλαμβανόταν στην αξιολόγηση συμμόρφωσης. Κανένας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για, τη δαπάνη, ε, για την ποιότητα των δαπανών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει αυτό δεν είναι πρόβλημα, αλλά των κρατών μελών. Και στο τέλο η απαλλαγή χορηγείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ξέρει ξεκάθαρα ποιο είναι υπεύθυνο γιατί. Ποιο επομίζεται τι ευθύνε. Και αν γίνει διακοπή και σταματήσει η χρηματοδότηση, πρέπει να είναι σαφέ ποιο έκανε το σφάλμα, ποιο είναι υπεύθυνο. Έτσι τα βλέπω εγώ. Λογικά, εγώ βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αποσυρθεί. Αλλά έχω την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως τελικά θέλει να είναι ξεκάθαρη η κατάσταση, να είναι ξεκάθαρο ποιος είναι υπεύθυνο και να μην κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα πάντα όσα κάνουν τα κράτη-μέλη. Και θέλει συγχρόνω τη διαδικασία να την κάνει πιο σύντομη, πιο βραχεία και πιο διαφανή. Ο ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ κατανοώ ότι υπήρξε μια σημαντική παράληψη στην αρχική μου παρέμβαση. Δεν ήθελα να μακρηγορήσω, αλλά δεν είπα τίποτα για το ρόλο της Κομισιόν. Είπα για το τι θα γίνει στα κράτη-μέλη, αλλά δεν ανέφερα τίποτα για το ρόλο της Κομισιόν. Πολύ σωστά αυτοί που έλαβαν το λόγο ανέφεραν ότι αυτό είναι ένα πολύ ζωτικό θέμα. Να υπογραμμίσω λοιπόν καταρχήν ότι δεν πρόκειται η Κομισιόν να υποβαθμίσει το ρόλο της ή όπως υπονοησμένοι να την κάνουν, να την κάνει και να αποσύσει την ευθύνη γιατί η Κομισιόν έχει μια ευθύνη βάσει των συνδικών που δεν μπορεί να αποδυναμωθεί. Δεύτερον, η Κομισιόν έχει αναπτύξει μια σαφή στρατηγική για το πώς θα πρέπει να φέρει σε πέρα στις ευθύνε της και θέλουμε να διατηρήσουμε αυτή τη στρατηγική. Ο τρόπος με τον οποίο εμείς θα εκπληρώνουμε τις ευθύνε μας είναι με την εφαρμογή της λεγόμενης προσέγγισης ενιαίας μορφής λογιστικού ελέγχου. Είδαμε αυτά τα χρόνια ότι δεν μπορεί η Κομισιόν να έχει την πρωτογενή ευθύνη για το λογιστικό έλεγχο διαφορετικών συστημάτων και εκατομμυρίων πράξεων στα κράτη-μέλη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βάση της ε, διαμοιρασμένης διαχείρισης είναι ακριβώς ευθύνη του κράτους μέλους να παρουσιάσει μια διακήρυξη αξιοπιστίας, η οποία πρέπει να παρουσιαστεί με κάποιο τρόπο, με μια ετήσια γνωμοδότηση λογιστικού ελέγχου και με την πιστοποίηση των αιτήσεων ε, για δαπάνε. Στο μέλλον θα καλύπτεται από μια ετήσια δήλωση διοικητικής διαχείρισης και με το πιστοποιητικό λογιστικού ελέγχου. Αλλά αυτά θα είναι τα στοιχεία από τα κράτη-μέλη για τις για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο η Κομισιόν δεν τα δέχεται αυτά με τα μάτια της ασφαλισμένα. Πρέπει να εξασφαλίσει ότι αυτές οι δηλώσεις πράγματι έχουν κάποια σχέση με την πραγματικότητα. Το κάνει αυτό με μια σειρά από δραστηριότητε που συμπεριλαμβάνουν λογιστικό έλεγχο, ο οποίος μπορεί να γίνει από την διεύθυνσή μας ελέγχου στα πλαίσια μιας ετήσιας στρατηγικής λογιστικού ελέγχου. Για την τρέχουσα περίοδο εμείς έχουμε εστιάσει την προσοχή μας στις αρχές ελέγχου, να εξασφαλίσουμε ότι το έργο τους είναι υψηλής ποιότητας, επομένως μας δίνει γνωμοδοτήσεις οι οποίες θα είναι αξιόπιστες. Και θα κάναμε και το ίδιο και με το νέο σύστημα το οποίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί, γιατί οι αρχές λογιστικού ελέγχου θα παίζουν ένα προεξάρχοντα ρόλο για να μπορούν να μας δίνουν και τις ε, γνωμοδοτήσεις λογιστικού ελέγχου. Αν μας ικανοποιεί λοιπόν η αρχή λογιστικού ελέγχου, και οι γνωμοδοτήσεις τους, τότε δεν είμαστε υποχρεωμένοι να επαναλάβουμε το έργο τους. Αυτό είναι σημαντικό σε σχέση με τους τελικούς αποδέκτες, οι οποίοι δεν θέλουν να έχουν μια σειρά, <clears throat> μια πληθώρα από ελεγκτές που έρχονται και ελέγχουν τις δράσεις τους. Ουσιαστικά λοιπόν ο ρόλος της Κομισιόν δεν θα αλλάξει. Το ένα στοιχείο το οποίο απλώς θέλω να αναφέρω, που είναι ακόμα ανοιχτή ανοιχτό το θέμα για τον ρόλο της Κομισιόν είναι η εκκίνηση αυτού του συστήματος. <clears throat> Γιατί για το σύστημα 2007-2013 η Κομισιόν ήταν απόλυτα εμπεπλεγμένη εφόσον για κάθε πρόγραμμα θα πρέπει να δώσουμε τα σχόλιά μας και να πούμε τελικά κατά πόσο αποδεχόμαστε ότι μπορούμε να δώσουμε το πράσινο φως ή όχι. Μέχρι ότου δίναμε το πράσινο φως δεν μπορούσαν να γίνουν καθόλου προκαταβολές ή ενδιάμεσες πληρωμές στα κράτη-μέλη. Ήταν λοιπόν ότι ανοίγει η βρύση μονάχα όταν η Κομισιόν ήταν ικανοποιημένη για την σωστή εκκίνηση των προγραμμάτων. Τώρα, βλέποντας πώς έχει λειτουργήσει το σύστημα στο παρελθόν και πώς μπορεί να λειτουργήσει το νέο σύστημα στο μέλλον, θα έχουμε τη διαδικασία διαπίστευσης που θα βασίζεται στην επιλογή του φορέα, του πιστοποιημένου φορέα και αυτό θα σημαίνει ότι δεν θα χρειάζεται για κάθε διαδικασία πιστοποίησης να ακολουθούμε την ίδια διαδικασία ελέγχου. Να έχουμε μια διαδικασία που, που θα είναι πιο εστιασμένη στον κίνδυνο. Να έχουμε λοιπόν την, ε, τον έλεγχο της διαπίστευσης στην αρχή και αν υπάρχουν προγράμματα τα οποία είχαν υψηλά κονδύλια και όχι περιορισμένα κονδύλια, να εστιάσουμε εκεί την προσοχή μας και επίσης σε όλους τους τομείς όπου από την τρέχουσα εμπειρία μας έχουμε κάποιες αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα και την επάρκεια του συστήματος. Πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τους πόρους μας και τα κράτη-μέλη επίσης. Δηλαδή εισάγουμε και ένα στοιχείο, αν θέλετε, αναλογικότητας σε ό,τι αφορά την προσαρμογή του ελέγχου, της προσπάθειας ελέγχου στους κινδύνους οι οποίοι υπάρχουν. Αλλά δεν πρόκειται η Κομισιόν να μειώσει το ρόλο της, να εκχωρήσει τις ευθύνες της ή οτιδήποτε τέτοιο. Μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο θα ενισχύσει τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη δίδουν τις εγγυήσει που απαιτεί η Κομισιόν και αυτό σημαίνει ότι αν τα πράγματα πηγαίνουν καλά και αν η Κομισιόν παίρνει στερεά στοιχεία κάθε χρόνο τα οποία δείχνουν ότι λειτουργεί το σύστημα θα μπορούσαμε στη συνέχεια να συμφωνήσουμε με το κράτος μέλος ότι πρώτον η Κομισιόν δεν θα χρειαζόταν να κάνει η ίδια πια λογιστικούς ελέγχους και θα μπορούσαμε να επιτύχουμε και μια αντίστοιχη μείωση στον ελεκτικό ρόλο του κράτους μέλους. Δεν θα θέλαμε να έχουμε υπερβολικό έλεγχο. Το επίπεδο ελέγχου θα πρέπει να είναι σύμμορφο με το επίπεδο κινδύνου. Και με τον τρόπο αυτό, με την ετήσια διαδικασία ελέγχου, θα μπορούσαμε να έχουμε εργαλεία που θα μας έδινε δυνατότητα να έχουμε μια πιο αναλογική αντιμετώπιση για τις απαιτήσει λογιστικού ελέγχου. Ας ξαναγυρίσω τώρα στα συγκεκριμένα σημεία τα οποία αναφέρθηκαν κατά τη συζήτηση από την πρόεδρό σας για την εδαφική συνεργασία καταρχήν για το 2013 και επέκεινα υπάρχουν ειδικοί κανόνες μας, πάντα θα υπάρχουν κάποιες ειδικές ρυθμίσεις Έχουμε ένα σύστημα με πολλά κράτη-μέλη τα οποία έχουν κοινά προγράμματα και υπάρχει μια διαχειριστική αρχή σε ένα κράτο μέλος και η αρχή λογιστικού ελέγχου κανονικά στο ίδιο κράτο μέλος. Αλλά οι φορείς αυτοί δεν μπορούν να ταξιδεύουν σε άλλα κράτη-μέλη για να κάνουν μόνοι του ελέγχου. Θα πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία εκχώρηση αρμοδιοτήτων και αυτό θα παραμείνει στο νέο σύστημα. Δεν θεωρούμε όμως ότι θα υπάρχουν θεμελιώδεις δυσκολίε για να εφαρμόσουμε αυτές τις αλλαγές. Και κατά κάποιο τρόπο η εξάλληψη της αρχής πιστοποίησης, της πιστοποιημένης αρχής, θα διευκολύνει αυτά τα διαμεθοριακά προγράμματα. Πιστεύουμε ότι έτσι θα απλοποιηθούν αυτές οι διαδικασίες. Το μόνο ερώτημα το οποίο θα πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι η διατύπωση μιας ετήσιας διαχειριστικής αρχής για μια αρχή που έχει να κάνει με ένα, ένα πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας γιατί δεν μπορούν να αναλάβουν την πλήρη ευθύνη για αυτά που γίνονται σε άλλα κράτη-μέλη έχουν βασίζονται στις δηλώσεις που έχουν δοθεί σε αυτά. Είναι λοιπόν μια πιο καταρακτικού χαρακτήρα διαδικασία όπου οι εθνικές αρχές δίδουν την αξιολόγησή τους για το τακτικό και το νόμιμο των ε, πράξεων αυτών των ε, ε, δαπανών και η διαχειριστική αρχή ελέγχει την πληρότητα και επιβεβαιώνει τα στοιχεία που δίνουν οι επιμέρους εθνικές αρχές. Σε επίπεδο όμως αρχιτεκτονικής, εμείς δεν βλέπουμε το θέμα αυτό τόσο προβληματικό. Νομίζω λοιπόν ότι έχω απαντήσει και στα άλλα ερωτήματα που έχουν να κάνουν με την αξιολόγηση συμμόρφωσης. Η κύρια αλλαγή είναι ότι η συμμόρφωση θα καλύπτει όλο το σύστημα, αλλά η διαπίστευτη θα είναι πιο εστιασμένη στον υποδιαπίστευση φορέα. Και η Κομισιόν θα παρεμβαίνει μονάχα σε περιπτώσεις που θεωρεί επικίνδυνες και θα εμπλεκόμαστε ήδη από την αρχή όπως κάνουμε τώρα με την ε, αξιολόγηση συμμόρφωσης. Εν πάση περιπτώσει, η Κομισιόν θα ξεκινούσε στην αρχή της προγραμματικής περίοδου και θα ακολουθούσε μια προσέγγιση επί τη βάση του εκτιμόμενου κινδύνου. Με στόχο να είμαστε σίγουροι ότι όλα αυτά τα οποία έχουν διατυπωθεί σε επίπεδο διαπίστευσης αντανακλούν την πραγματικότητα σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των κριτηρίων πιστοποίησης. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο θέλουμε να έχουμε μια προσέγγιση περισσότερο από τη βάση κινδύνου. Γιατί για την ε, αξιολόγηση συμμόρφωσης αυτό ήταν ένα πάρα πολύ τιτάνιο έργο για την Κομισιόν, καταδαπανούσε πάρα πολλούς πόρους και μας εμπόδιζε να κάνουμε άλλα πράγματα συγχρόνως. Αν λοιπόν υπάρξει μια πιο αναλογική εμπλοκή της Κομισιόν στα θέματα αυτά, μπορούμε να ξεκινήσουμε τα προγράμματα πιο γρήγορα, κάτι το οποίο είναι πολύ πιο σημαντικό και να εστιάσουμε την προσοχή μας στις περιοχές υψηλού κινδύνου. Για να επανέλθω σε μερικά ακόμα στοιχεία τα οποία αναφέρθηκαν. Το ετήσιο έτος της καταγραφής. Είναι πολύ δύσκολο να σας το εξηγήσω χωρίς να έχω διαγράμματα. Θα έπρεπε να έχω ένα διάγραμμα να σας δείξω πώς εκτελήσονται τα πράγματα στον χρόνο. Στην πολιτική μας όμως <clears throat> υπάρχει μια χρονική υστέρηση μεταξύ της στιγμής που γίνεται η πραγματική καταβολή των χρημάτων προς ένα δικαιούχο και η επιστροφή στα κράτη-μέλη ή στον δικαιούχο από την Κομισιόν. Γιατί όταν γίνεται η δαπάνη δηλώνεται και ελέγχεται και μετά η Κομισιόν καταβάλει το αντίστοιχο ποσό. Υπάρχει λοιπόν μια σειρά δράσεων προτού έρθει μια δαπάνη στην Κομισιόν και ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφής των εξόδων. Αν πάρετε λοιπόν ένα χρόνο μέσα στον προπολογισμό της Κομισιόν, έχετε ένα σύνολο από επιστροφέ που εκταμιεύονται από την Κομισιόν στα κράτη-μέλη. Αν όμω θέλετε να συνδέσετε αυτό με τι δαπάνε οι οποίε γίνονται από του τελικού αποδέκτε στα κράτη-μέλη, θα πρέπει να πάτε λιγάκι στο παρελθόν. Γιατί δεν είναι το ίδιο οικονομικό έτος που συνδέεται με αυτές τις δαπάνες. Το να έχουμε λοιπόν μια οριακή <clears throat> ημερομηνία για το έτος λογιστικής, μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη αντιστοιχία. Σταματάει το έτος λογιστικής στις 30 Σεπτεμβρίου, οπότε οι, αρχε... οι πληρωμές που έχουν γίνει από τις εθνικές αρχές στους δικαιούχους θα μπορεί λοιπόν η Κομισιόν να ελέγχει μονάχα τις ε, πληρωμές που έχουν γίνει μετά από έλεγχο σε, στα κράτη-μέλη. Και έτσι θα έχουμε πλήρη αντιστοιχεία αυτών που πληρώνουμε εμείς σε ένα οικονομικό έτος και αυτών που μας έχουν ζητηθεί από τα κράτη-μέλη. Έτσι λοιπόν αν έχουμε μία σχέση του έτους λογιστικής απεικόνησης με το οικονομικό έτος, τα, οι δύο καταγραφές αντιστοιχούν, έχουν ακριβώς τις ίδιες δαπάνες που έχουμε καλύψει εμείς σε ένα οικονομικό έτος. Αυτό διευκολύνει τα μάλα την διαδικασία ε, εκαθάρισης και απαλλαγής. Βέβαια δεν αλλάζει το δικό μας οικονομικό έτος και τη διαδικασία απαλλαγής εκτός από μια θετική επίπτωση ότι μας επιτρέψει σε επίπεδο απαλλαγής να δείξουμε πώς εμείς μπορούμε να καταλήξουμε σε μια εξασφάλιση από τους ελέγχους που έχουν γίνει επιτοπίως από τις ελεγκτικές αρχές ότι τα πράγματα είναι εντάξει, ότι έχουν γίνει δαπάνες με νομότυπο και επακριβή τρόπο. Προς το παρόν δεν μπορούμε εμείς να καταδείξουμε πλήρως την αντιστοιχία μεταξύ των χρηματοδοτήσεών μας και των δαπανών που γίνονται επιτοπίως. Κάτι ακόμα για το ρόλο της Κομισιόν και την ανάγκη να ενισχύσουμε το ρόλο της Κομισιόν. Ένα σημείο που δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή με το νέο δημοσιονομικό κανονισμό, ένα από του κύριου τρόπου με του οποίου εμεί έχουμε ενισχύσει το ρόλο τη Κομισιόν για το 2013, είναι με την δυνατότητα να αναστείλουμε τις ε, πληρωμές όταν υπάρχουν στοιχεία ότι το σύστημα έχει αδυναμίες. Θέλουμε να το διατηρήσουμε λοιπόν αυτό το στοιχείο γιατί αυτό ακριβώς μας επιτρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στα μαύρα πρόβατα και στους μαύρους κύκνους, εκεί που τα κράτη-μέλη έχουν προβλήματα να μπορέσουν να εφαρμόσουν αποτελεσματικά συστήματα. Πιστεύω λοιπόν από τη μία πλευρά θα διατηρήσουμε αυτή τη δυνατότητα να διακόπτουμε και να αναστέλουμε τις πληρώμες για τα προγράμματα αυτά όπου φάνηκε να υπάρχουν κάποιες αδυναμίες και ελλείψεις, αλλά από την άλλη πλευρά ενισχύουμε το σύστημα δίνοντα τα κράτη-μέλη την υπευθυνότητα να αποδιαπιστεύσει, να άρει τη διαπίστευση των φορέων αυτών όταν δεν έχουν λειτουργήσει σωστά, όταν φαίνεται ότι η διαχειριστική αρχή δεν έχει επιτύχει αυτά τα οποία έπρεπε να επιτύχει, ότι δεν έχει την ικανότητα ή οτιδήποτε άλλο για να δώσει μια σωστή διαχείριση και ένα σωστό έλεγχο, τότε το κράτος μέλος δεν έχει καμία υποχρέωση να πάρει αυτή την ε, ε, διαπίστευση και να τη δώσει σε κάποιο άλλο φορέα. Το να υπάρχει η υποχρέωση όταν υπάρχει ένα πρόβλημα να αποσυρθεί η διαπίστευση, αυτό υπευθυνοποιεί το κράτο μέλο για να μπορεί να πει ότι είτε αυτοί οι φορεί έχουν την απαραίτητη δεξιότητα, προσόντα, προσωπικό κτλ. ή αλλιώ δεν έχουν τη διαπίστευση και τότε τα κράτη-μέλη πρέπει να βρουν κάποιον άλλο φορέα που θα αναλάβει αυτή την ευθύνη, αλλιώ δεν πρόκειται να έρθει καθόλου χρήμα από την Κομισιόν. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και το τελευταίο σημείο το οποίο θα δείξω σε σχέση με τις περιφέρειες. Όλα αυτά που σας είπα σε επίπεδο συστημάτων, αυτά και εξαρτάται από την θεσμική αρχιτεκτονική των κρατών μελών και πώς λειτουργεί η διακυβέρνηση σε πολλά επίπεδα, όλα αυτά μπορούν να γίνουν σε εθνικό επίπεδο ή σε περιφερειακό επίπεδο, ίσως σε ορισμένα κράτη-μέλη. Όταν μιλάμε για μια διαπιστευτική αρχή, ένα φορέα πιστοποίηση, αυτός ο φορέας μπορεί να είναι σε περιφερειακό επίπεδο. Υπάρχουν πάρα πολλές λοιπόν παραλλαγές οι οποίες μπορούν να ισχύουν, είτε μια αρχή για όλο το κράτος αλλά με πολλούς διαπιστευμένους φορείς, είτε μια αρχή διαπίστευσης ανά περιφέρεια και ένα διαπιστευμένο φορέα ανά περιφέρεια. Δεν υπάρχει λοιπόν εδώ πέρα μονάχα μία λύση, αυτό εξαρτάται από τις θεσμικές λύσεις που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτό το σημείο. Τις επόμενες εβδομάδες, Γιάν, θα εργαστούμε επί τη βάση της υποθέσεως ότι η ψηφοφορία στην καθήλυνα αρμόδια επιτροπή θα δεξαχθεί τον Ιούνιο, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά την ημερομηνία του Ιουνίου. Δεν ξέρουμε ακόμα όμω, πρέπει να υποθέσουμε ότι θα πρέπει το σχέδιο γνωμοδότηση να το έχουμε έτοιμο για τον Απρίλιο για την Ρέτζη Αν αναβληθεί και αλλάξει ημερομηνία, θα προσαρμόσουμε δεόντω το χρονοδιάγραμμα. Όσοι θέλουν να συνεργαστούν με τον εισηγητή στενότερα είναι πρόσδεκτοι. Ας το κάνετε τώρα και δεν χρειάζεται να περιμένετε για την περίοδο υποβολής τροπολογιών. Γιάν, ένα σχόλιο απευθυνό Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ίσως φάλω, αλλά έχω την εντύπωση ότι ανοίγετε τους ασκούστε όλου με τον αριθμό των ε, φορέων που μπορούν να χορηγήσουν διαπιστεύσεις, εγκρίσεις. Και εξηγήστε το στο μέλλον. Είπατε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερους φορείς διαπίστευσης. Εκεί γεννάται άλλο ζήτημα. Είναι ξεκάθαρο να λέμε ένας φορέας κατά χώρα και αλλά είπατε ε, ένα ομόσπονδο κρατήδιο σε ομόσπονδη χώρα, αλλά είπατε μετά είναι και ενδεχόμενο να υπάρχει ένα φορέα για κάθε περιφέρεια. Αυτό είναι πολύ παρακινδυνευμένο. Δεν το σου Αυτό είναι ένα σχόλιο. Πρόεδρο, να εξηγήσω του συναδέλφου. Ο Λαμπέρ έχει το λόγο. Στο δικό μου ερώτημα για τη θέση της Επιτροπής Ρέτζι όσον αφορά τους κανονισμούς που να θεσπίσουμε αργότερα. Καλό θα ήταν να καλέσουμε τον εισηγητή που είναι στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού και ασχολείται με το θέμα να έρθει εδώ και να το κουβεντιάσουμε. Διότι θα πρέπει να γίνει άμεσα, απευθεία αυτή η συζήτηση, πιστεύω. Αυτό θα πρότεινα. Εγώ θα πρότεινα το εξή, λέει ο Πρόεδρο. Αυτό ο δημοσιονομικό κανονισμό είναι σημαντικότατο για την μελλοντική πολιτική συνοχή. Διότι όταν ψηφιστεί και εγκριθεί και υιοθετηθεί και εφαρμοστεί θα έχει αντίκτυπο και στον κανονισμό για την πολιτική συνοχής που θα διαπραγματευτούμε τον επόμενο χρόνο. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να συζητήσουμε εκτενώς το θέμα. Γι' αυτό θα ήθελα να προτείνω το εξής. Μήπως στα πλαίσια της Επιτροπής που έχουμε φορτωμένο πρόγραμμα πριν το θέρος, διοργανώσουμε έκτακτη σύνοδο για εκείνους που θέλουν να συμμετάσχουν, να καλέσουμε τους εισηγητές της Επιτροπής Προϋπολογισμών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ίσως αν θέλω να είμαι κακή και κάποια κράτη-μέλη, ούτως ώστε να καταλάβουμε άριστα το τι αποφασίζουμε. Να καταλάβουμε, όχι να είμαστε αντίθετοι, να καταλάβουμε. Ε, διότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για τις συζητήσεις μας για το δημοσιονομικό κανονισμό. Ελπίζω να είστε όλοι έτοιμοι να συνεργαστείτε και πιθανότατα θα συνεχίσουμε, Γιάν, υπό την προεδρία σου τη συζήτηση για τον κανονισμό αυτόν. Ευχαριστώ όλους πάρα πολύ, κυρίως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζουμε να διαβιβάσετε τα σχόλια και τις αμφιβολίες που εκφράσαμε στους αρμοδίους το λάβετε υπόψη στι περαιτέρω εργασίε σα και να λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη σα τη διαφορά μεταξύ κοινή αγροτική πολιτική και τη πολιτική συνοχή και το πώ λειτουργούν. Με αυτό σα ευχαριστώ και προχωρώ στο επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη. Η έκθεση Σαμπίν Βερχάιν Ευρωπαϊκά Δίκτυα Ευρυζωνικότητα. Και μετά από τη Σαμπίν θα ζητήσω από τους σκιώδεις να είναι έτοιμοι αν θέλουν να προσθέσουν κάτι. Η Σαμπίν έχει το λόγο. Πρόεδρε, συνάδελφοι, να ευχαριστήσω καταρχάς τους Κιώδης για την καλή συνεργασία. Πρωτού περάσω στα μεμονωμένα ζητήματα στην γνωματοδότηση, θα ήθελα να υποδείξω ότι υπήρξαν κάποιες, κάποια προβλήματα στην παράγραφο 4 και 5 σε ό,τι αφορά τη μετάφραση έχουν βελτιωθεί, έχουν ε, διορθωθεί τα λάθη. Αυτά από όσο ξέρω στην αγγλική εκδοχή του κειμένου, δεν μπορούσα φυσικά να το ελέγξω σε όλες τις γλωσσικές εκδοχές, αλλά υπήρξε μία σύγχυση, νομίζω ότι θα διευκρινιστεί όμως. Στη γνωμοδέτηση, ναι, μα συγγνώμη, λέει η πρόεδρο, διακόπτη σα, παρακαλώ συνάδελφοι. Όσοι θέλουν να φύγουν, α φύγουν, αλλά σα παρακαλούμε με απόλυτη ησυχία. Η κυρία Ευχαριστώ. Προσπάθησα λοιπόν να κοιτάξω την πλευρά της περιφερειακής ε, ανάπτυξης σε ό,τι αφορά τα δίκτυα ευρυζωνικότητας και επικεντρώθηκα σε κάποια περιορισμένα θέματα γιατί μας ε, περιορίζουν και σε ό,τι αφορά τους χαρακτήρες πλέον στην ε, γνωμοδότηση. Ελπίζω να λάβω τροπολογίες και έτσι να εμπλουτίσουμε την γνωμοδότηση, να σας παρουσιάσω ποια είναι τα βασικά ζητήματα όμως. Καταρχάς πρόκειται για μια βασική αξίωση προκειμένου να αναγνωριστεί η βριζονική ε, παροχή ως βασική υπηρεσία. Δεν μπορούμε να μην έχουμε πρόσβαση σε ίντερνετ αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στην Ευρώπη και το πρόβλημα είναι ότι στην Ήπεθρον η αγορά έχει εν μέρη αποτύχει γιατί είναι περιορισμένοι οι κάτοικοι και άρα οι ενδυνάμοι πελάτες και φυσικά αυτό δεν παρέχει κίνητρα για να επιταχυνθεί η υπερτερό ανάπτυξη των δικτύων ευρυζωνικότητας και αυτό τι σημαίνει ότι υπάρχει μείωση και του ενδιαφέροντος και δεν υπάρχει τόσο ελκυστικός χαρακτήρας στην ύπεθρο σε ό,τι αφορά τον οικονομικό χαρακτήρα δηλαδή, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις. Κοιτώντας τα θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ε, και αν θέλουμε να ε, ενισχύσουμε και να προωθήσουμε τέτοια προγράμματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής εκμάθησης και το καθεξής, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ευρυζωνικής ε, ε, ε παροχής. Θα πρέπει λοιπόν το συντομότερο δυνατόν να είναι απόλυτη η κάλυψη της βασικής αυτής υπηρεσίας για να μην υπάρχει και αποκοπή από τις άλλες περιφόρειες. Είναι θέμα βασικό, όπως και το νερό, ο ηλεκτρισμός και νομίζω ότι θα συνδράμει και στην ε, εξίσωση των όρων διαβίωσης. Δεύτερο στοιχείο αναφέρομαι στις διαδικασίες και στα προγράμματα ενίσχυσης. Θεωρώ ότι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να υπάρχει απλοποίηση των προγραμμάτων και των διαδικασιών προκειμένου να είναι αποδοτική και γρήγορη η παροχή των ενισχύσεων, η ροή των πιστώσεων. Και επίσης να, υπάρχει, να υπάρχουν διάφορες φάσεις σε κάθε πρόγραμμα. Καλώ ορίζω λοιπόν ε, την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την... να διατηθούν τέτοιες υπηρεσίες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί θεωρώ ότι τα προγράμματα σύμπραξης μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα μπορούν να οδηγήσουν σε επιτυχίες στην Ήπεθρο, όπου ε, για οικονομικούς λόγους ίσως να μην αξίζει τον κόπο να δραστηριοποιηθεί μια επιχείρηση. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στις τοπικές και περιφερειακές ε, αρχές να καταστήσουν το περιβάλλον πιο, πιο ελκυστικό για τις ε, επιχειρήσεις. Γιατί μεγάλο τμήμα των, ε, του κόστους και των δαπανών προέρχεται από την, την κατασκευή των υποδομών και όλα αυτά μπορούν να βαλτιστοποιηθούν. Θα πρέπει να αναπτυχθούν και καινούργια συστήματα για συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Τρίτο το σημείο. Αναφέρομαι στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Παρενισχύσεων, η οποία θα πρέπει να απλουστευτεί. Οι προδιαγραφές θα πρέπει να απλουστευτούν είναι αντικειμενικές, είναι αντικειμενικά τα κριτήρια που προβλέπονται και στα πλαίσια των ε, τελευταίων μεταρρυθμίσεων απλοποιήθηκαν και για την ευρυζωνικότητα, αλλά εξακολουθεί να είναι επαχθές το σύστημα για την διοικητική εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών και δεν είναι δυνατόν ε, τέτοιες δαπάνες ευρωπαϊκές να καταλήγουν στα ταμεία ιδιωτικών εταιριών σε μεγάλο βαθμό. Γιατί θεωρούμε ότι στην παρούσα φάση μεγάλο τμήμα των χρημάτων δαπανάται για γνωμοδοτήσεις για τον σωστό τρόπο διαμόρφωσης συμπράξεων. Και η σημερινή κατάσταση οδηγεί σε νομική αβεβαιότητα στην πράξη εν μέρη σήμερα. Και αυτό φυσικά έχει τον αντίκτυπό του και για τις επενδύσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει πώς μπορεί να διαμορφωθεί με πιο φιλικό για τι επενδύσεις τρόπο το σύστημα. Θα πρέπει στο πλαίσιο αυτό να σκεφτούμε κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχει ίσως ε, σε ό,τι αφορά την ε, νομοθεσία περί ενισχύσεων ε, μία πρόβλεψη για απαλλαγή σε περίπτωση ε, περίπλοκο, περίπλοκων μονομένων διαδικασιών. Ίσως να υπάρχουν κάποια τυποποιημένα συστήματα. Τέταρτο σημείο αναφέρομαι στην ε, καθολική παροχή τέτοιων δικτύων. Αναφέρομαι σε προγράμματα όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εξαποστάσεως εκμάθηση που αφορούν και μικρομεσαίες επιχειρησίες. Στην Ήπεθρο οι επιχειρήσεις δεν χρειάζονται μόνο μια διαρκή τέτοια δυνατότητα και ικανότητα, αλλά να έχουν και δυνατότητα να ανεβάζουν, για παράδειγμα, ε, με ταχύες, ε, ταχύτητες ε, πληροφορίες και δεν αρκούν πάντα οι δυνατότητες που υπάρχουν προκειμένου δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τέτοια ε, ταχαία δίκτυα. Και υπάρχουν κάποιες τεχνολογίες ε, γέφυρας, αν θέλετε. Δεν αρκεί σήμερα η τεχνολογία για να παρέχεται ευρυζωνικότητα διαρκώς. Και εδώ λοιπόν θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε κινητές ε, τεχνολογίες, οι οποίες όμως δεν πρόκειται να γεφυρώσουν το ψηφιακό χάσμα που υπάρχει. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να επενδύσουμε προς αυτή την κατεύθυνση σε ε, υποδομής, για παράδειγμα. Να υπάρχει μια φάση εκπαίδευσης προκειμένου να μπορέσουν και οι επιχειρήσεις να υποφεληθούν μελλοντικά από το σύστημα αυτό και στην Ήπεθρο. Θα πρέπει να, να ενισχυθούν οι οπτικές ίνες γυαλιού και νομίζω ότι αυτή η τεχνολογία που χρηματοδοτείται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί πλέον να λείπει σε καμία περίπτωση. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η τεχνολογία των ε, οπτικών ινών είναι η τεχνολογία επιλογής μας και θα πρέπει να την ε, προτιμήσουμε. γιατί έτσι θα αναπτυχθεί πλήρως το δυναμικό ανάπτυξης και έτσι θα αυξηθεί και η ποσότητα δεδομένων για το μέλλον. Ελπίζω λοιπόν να λάβω πολλές παρατηρήσεις από πλευρά σας, πολλές προσθήκες και χαίρομαι και για τη μελλοντική καλή συνεργασία με τους κοιότης και με τους υπόλοιπους ε, συναδέλφους από την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τόιρερ. Ευχαριστώ. Τον Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτό το σχέδιο γνωμοδότηση. Νομίζω ότι έχουμε μια πολύ καλή παρουσίαση των αναγκών για την ε, τροφοδοσία σε ευζωνικά δίκτυα που είναι και η αχίλιος πτέρνα της ε, κατά κάποιο τρόπο κοινωνίας της πληροφόρησης στην Ευρώπη υπάρχουν πολλές φορές ε, γραφεία δικηγορικά ή γραφεία αρχιτεκτονικά ή ακόμα και οι ιατροί οι οποίοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν σωστά σε απομονωμένες περιοχές γιατί δεν έχουν αρκετή ε, παροχή ευρυζωνικών δεδομένων. Επομένως όλα αυτά τα οποία λέμε για την κοινωνία της πληροφόρησης έρχονται σε αμφιβολία, τίθεται σε αμφιβολία αν δεν μπορεί να λειτουργήσει η πρόσβαση στα ευρυζωνικά δίκτυα. Είναι απαραίτητο λοιπόν να έχουν όλοι πρόσβαση σε αυτή την τεχνολογία. Αυτό είναι μια βασική απέτηση και πρέπει να εξασφαλιστεί επομένω. Επίσης, τα λέει η ανακοίνωση της Κομισιόν ότι δεν υπήρξε επαρκής απορρόφηση των μέσων που έχουν τεθεί σε διάθεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να ξέρω και εγώ γιατί δεν έχει γίνει αυτή η απορρόφηση από τη γερμανική πλευρά. Μπορώ να φανταστώ ότι σε πολλές, ε, σε πολλές ε, περιοχές, σε πολλούς δήμους λένε ότι δεν θέλουν να επενδύσουν τόσα πολλά χρήματα στο να έχουν μία ε, ευ, μια τεχνολογία η οποία να είναι ασύρματου χαρακτήρα. Δεν ξέρω λοιπόν αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ακολουθήσει μια πιο ουδέτερη ως προς την τεχνολογία αντιμετώπιση ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν επίγεια και υπόγεια δίκτυα ευρυζωνικά παραγωγικά με οπτικές ίνες κτλ οι περιοχές αυτές. Κάτι ακόμα για να, εφόσον βρισκόμαστε ακόμα στην πρώτη αυτή ανταλλαγή απόψεων, αν δεν ε, αποκλείσει κανείς τελείως την ε, δυνατότητα να υπάρχει τεχνολογία ευρυζωνική μέσω ασύρματων δικτύων, δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε τη δυνατότητα το τελευταίο μίλι, το λεγόμενο τελευταίο μίλι, δηλαδή η σύνδεση με τον καταναλωτή, να γίνεται με επίγεια δίκτυα. Υπάρχει το θέμα λοιπόν όχι μόνο το ότι τα σύρματα δίκτυα έχουν λιγότερη δυνατότητα ε, μετάδοσης πληροφοριών αλλά και το λεγόμενο ηλεκτρονικό smog δηλαδή η μεγάλη, ε, ο μεγάλος θόρυβος, οι μεγάλες παρεμβολές οι οποίες μπορούν να προκύψουν στα σύρματα δίκτυα. Πρέπει λοιπόν και πολλές φορές και για λόγους ε, κινδύνου στην ε, ανθρώπινη υγεία να αποκλείσουμε τις δυνατότητες αυτές να υπάρχουν ασύρματα δίκτυα για το, τα ευρυζωνικά. Η Έλισσα Πετσφέντερ θα σας ευχαριστήσω και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια η οποία κατά την άποψή μας έχει καταφέρει να παρουσιάσει τα ουσιώδη και εγώ υποστηρίζω απόλυτα αυτά τα οποία λέει ότι ουσιαστικά θέτουμε σε αποκλεισμό τις περιοχές οι οποίες δεν έχουν την πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα και αυτό είναι μια ουσιαστική, ένα ουσιαστικό πρόβλημα και σε ορισμένες περιοχές τη Αγγλία και τη Γερμανία, μερικοί νομίζουν ότι είναι 20 χρόνια στο παρελθόν γιατί δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δίκτυα. Περιοχέ οι οποίε είναι βέβαια αραιοκατοκιμένες, θα πρέπει να εξασφαλίσει αυτή η ευρυζωνική πρόσβαση με ασύρματα δίκτυα. Το ουσιαστικό είναι να τονίσουμε ότι αυτή η υπηρεσία πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια οικουμενική υπηρεσία, η πρόσβαση στα ευρυζωνικά δίκτυα και συμμερίζομαι αυτό το οποίο είπε και ο κύριος Τόιερ, ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι γίνεται η καλή χρηματοδότηση και για πιο ε, αηφόρες λύσεις. Τώρα, αν είναι καλύτερη η ασύρματη η ασύρματη λύση, δηλαδή με ραδιοφωνικά δίκτυα ή η λύση με επίγεια και υπόγεια καλώθια, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε σε κάθε περίπτωση. Ξέρω ότι γνωρίζετε το πρόβλημα αυτό, ότι ακόμα και στην περιφέρεια του Βερολίνου δεν είναι δεδομένο ότι μπορεί να έχει κανείς τη σωστή ευζωνική σύνδεση γιατί οι πάροχοι θεωρούν ότι ορισμένε περιοχέ μπορεί να μην είναι επικερδείς για να τους δώσουν καλύτερη υπηρεσία. Και όταν θέλουμε να δώσουμε δημόσια χρήματα για μια τέτοια λύση είναι φανερό ότι πρέπει να υπάρχει οικουμενικός χαρακτήρας στην υπηρεσία αυτή και θα πρέπει επίσης να σκεφτούμε μήπως η λύση που ακολουθούμε είναι η πιο πολύ δάπανη. να μην καταλήξει ο καταναλωτής λόγω της οικουμενικής υπηρεσίας να πληρώνει περισσότερο από ότι ορισμένοι άλλοι. Πρέπει να τονίσουμε λοιπόν και την οικουμενικότητα, αλλά και το να είναι οι σωστές οι λύσεις οι οποίες θα ακολουθηθούν και ίσως και με τις τροπολογίες μας μπορούμε να το τονίσουμε αυτό ακόμα περισσότερο ότι θα πρέπει να εξετάσουμε σε ποιο βαθμό ο πάροχος ο οποίος παίρνει μια δημόσια εντολή, ένα, μια δημόσια χρηματοδότηση για ένα δίκτυο, κατά πόσο είναι υπεύθυνο να εξασφαλίσει την ε, λειτουργία αυτού του δικτύου σε συνεργασία και με άλλες ε, μορφές ε, οικουμενικών υπηρεσιών σε περιοχές οι οποίες είναι αραιοκατοκυμένες. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε πολλές φορές σε περιοχές και όπου πρέπει να υπάρξουν σημαντικές τροποποιήσεις. Υπάρχουν περιοχές όπως η Σκοτία και η Ιρλανδία και στη Γερμανία έχουμε περιοχές αυτού του είδους. Και θα πρέπει να εξετάσουμε να εξασφαλίσουμε ότι όλες αυτές τις ε, μειονεκτικές περιοχές ε, ότι θα έχουν την κατάλληλη λύση και όχι να αφήσουμε αυτό το θέμα να το πάρει μια άλλη Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για μας στην Επιτροπή Περιφερειακών Θεμάτων, είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι οι περιοχές αυτές, οι οποίες είναι απομονωμένες ή αεροκατοικημένες, δεν θα βρεθούν σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τις άλλες περιοχές. Συνάδελφοι, έχουμε ακόμα τέσσερις ομιλητές για αυτό το θέμα και δύο γνωμοδοτήσεις για ενέργεια και γενή αγροτική πολιτική και πρέπει να συζητήσουμε και τις έξι. Παρακαλώ να περιορίζετε σε ένα λεπτό και θα τα καταφέρουμε. Ο κύριος Ντεάντζελης έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ καλή δουλειά που έκανε η συγγήτρια. Η ταχεία πρόσβαση, η υπερταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορεί να δώσει σημαντικότατη όθηση στην οικονομική ανάκαμψη. Κυρίως υπενθυμίστηκε, υπενθυμίστηκε αυτό ότι αυτό έχει σημασία για την Ήπεθρο. Είναι πολύ σημαντικές οι νέες τεχνολογίες και γι' αυτό το λόγο οι επενδύσεις σε νέα ανοιχτά δίκτυα κυρίως τα αγωνιστικά δίκτυα και μέσω της υποστήριξης του δημόσιου τομέα είναι η καλύτερη εγγύηση για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Θα ήθελα εντάχει να υπογραμμίσω κάποια σημεία που θεωρώ πρώτη της σημασίας για την ανάπτυξη του προγράμματος της ευρυζωνικής κυρίως όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και προσβασιμότητα στα νέα δίκτυα. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οι περιφέρειες χρειάζεται να ξεπεράσουν εμπόδια αλλά και καθυστερήσεις και μέσω ναι, μιας επένδυσης πολιτικής και οικονομικής όσον αφορά την καινοτομή τεχνολογική μπορεί να βοηθηθούν. Αλλά έχουμε στα τέσσερα ζητήματα και ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα να εξασφαλιστεί πρώτα απ' όλα ο ανταγωνισμό, υποστηρίζοντα την ανάπτυξη ανοιχτών αρχιτεκτονικών και να αποφύγει ο κίνδυνο μονοπωλίου όσον αφορά την αγορά. Δεύτερον, προσβασιμότητα ε, και από πλευρά των επενδυτών σε νέα δίκτυα με οπτική ίνα. Είναι ένα μέτρο θεωρείται αναγκαίο για να αποφευθεί η αύξηση του κόστους ε, των καλωδίων. Μετά τα τέλη για την πρόσβαση. Θα πρέπει να είναι δίκαια, ε, δίκαια τα τέλη. Θα πρέπει να εκμεταλλεύονται ανταγωνιστικέ υπηρεσίες ή καταναλωτές και όσον αφορά το κόστος. Θα πρέπει να εισαχθούν υπολογισμοί του κόστου κοινοί στα κράτη-μέλη για να προχωρήσουμε σε πιο ισότιμη βάση όσον αφορά τη διάδοση των νέων δικτύων. Και τέταρτον ερώτημα, και κλείνω εδώ, η ολική κάλυψη. Ουσιαστικά δεν πρέπει να μείνουν εκτός αναπτύξεως οι περιφέρειες της υπαίθρου, άρα χρειάζονται περισσότεροι πόροι για αυτές τις περιφέρειες, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν σε αυτό το τομέα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σον Κέλλη και παρακαλώ σύντομα. Θα είμαι σύντομο, θα είμαι σύντομο. Ευχαριστώ. Σαμπίν ε, Σόμερ αναφέρθηκε πολύ σωστά στο όλο θέμα και γενικότερα αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους του 2020 και να είναι ανταγωνιστική η Ευρώπη, κάτι που πρέπει να γίνει, τότε η ευρυζωνική είναι σημαντικότατη και για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν τεράστια κενά και δεν προχωράμε αρκετά γρήγορα και νομίζω ότι θα έχουμε πολλά κίνητρα να δημιουργηθούν ε, περισσότερες μικρομεσές, είναι καλό να, να είναι ανεξάρτητε από την. Οι μικρομεσαίε θα είναι ανεξάρτητε όσον αφορά τον τόπο εγκατάσταση, αν έχουν ευρυζωνική. Χωρί αυτή δεν έχουν την πρόσβαση. Μετά έχουμε την οδηγία για, για τι υπηρεσίε και για τα πνευματικά δικαιώματα. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά, αλλά δεν μπορούμε να πετύχουμε πλήρω του στόχου χωρί την ευρυζωνική. Το ίδιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονική υγεία κλπ και θα πρέπει να έχουμε ευρυζωνική τώρα, εξίσου σημαντικό όπω ε, να έχει κανεί και έναν δρόμο πάει στο σπίτι του. Τόσο σημαντική είναι η ευρυζωνική. Και όσο περισσότερου πόρου διαθέσουμε, τόσο καλύτερα θα μα δώσει καρπού βραχυπρόθεσμα. Ε, εδώ και δύο εβδομάδε θέλει να δώσει ευρυζωνική σε όλη τη χώρα μου στα πέντε χρόνια. Το είπα εσεί σε όλη την Ευρώπη. Εάν έχει όλη η Ευρώπη ευρυζωνική, Κυρίω η την επόμενη πενταετία ίσω να πετύχουμε τους στόχους του 2020, αδιαφορετικά δεν θα πετύχουμε τους στόχους χωρί στην Ευρυζωνική. Ευχαριστώ Σον, η κυρία Αντέλη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Εγώ να σας επιστήσω την προσοχή επί πραγματικού προβλήματος της δημόσιας υγείας. Ψηφιακά τα πάντα είναι καλά και άγια ευρυζωνική είναι πάρα πολύ καλή, αλλά υπάρχουν άτομα που δεν την αντέχουν. Είναι τα άτομα που έχουν ευαισθησία όσον αφορά την ηλεκτρονική τεχνολογία. Τι κάνουμε λοιπόν. Σε αυτή την έκθεση θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχει ένα, ένας όρος. Θα πούμε ότι θα εφαρμόσουμε την ευρυζωνική. Εκεί που μπορούμε να έχουμε ευρυζωνική, αν έχουμε τη συμφωνία των κατοίκων και των ενώσεων καταναλωτών κλπ. Έχουμε ένα καθήκον να ζητήσουμε την άποψή τους. Νομίζω ότι είναι πραγματικά χρήσιμο αυτό και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λαμπέρ Φανίστελροϊ. Πρόεδρε, καταλαβαίνω και εγώ τη συμμετοχή της περιφερειακής διάστασης. Κάποιες τροπολογίες να διατυπώσω. Συζητήσαμε ως αρχή της περιφερειακής ε, πολιτικής και της εδαφικής διάστασης και είπαμε ότι είναι πολύ καλό να υπάρχει ε, επικέντρωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την έρευνα, για την τεχνολογία. Φυσικά θα πρέπει να το κάνουμε αυτό για να είμαστε ανταγωνιστικοί και καλύτεροι σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε όλο τον κόσμο. Αυτό γίνεται μόνο με συνεργασία και σύνδεση. Και αυτό αναφέρθηκε στο, στην πράσινο βίβλο για την εδαφική ε, συνεργασία. Χρειαζόμαστε λοιπόν συγκέντρωση, συνεργασία και σύνδεση, τα τρία C's. Χρειαζόμαστε λοιπόν ευρυζωνικότητα. Και θα ήθελα αυτό κάπου να μπει στο κείμενο. Κατά δεύτερον, σε ό,τι αφορά τις απτικές ίνες ε, γυαλιού. Πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Αλλά η περαιτέρω συμπλήρωση με τεχνολογίες δορυφορικές θα είναι απαραίτητε και θα πρέπει να συνεχίζονται μάλλον και οι εξελίξει αυτέ. Θα πρέπει να είμαστε ουδέτεροι από πλευρά τεχνολογία, από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί μπορεί σε 5-10 χρόνια να έχουν προκύψει τεχνολογίε τι οποίε δεν φανταζόμαστε καν σήμερα. Thank you, Ευχαριστώ, Λαμπέρ. Σαμπίν, έχει κάτι να προσθέσει. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά τα οποία έχετε προσθέσει στη συζήτηση και στην αρχική μου πρόταση αναφέρονταν και η δορυφορική τεχνολογία για λόγους έλλειψης χώρου χρειάστηκε να μην το αναφέρω. Σίγουρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλες τις υπάρχουσες τεχνολογίες για να μπορέσουμε να δώσουμε σε όλους, σε όλες τις περιοχές την απαραίτητη πρόσβαση σε γρήγορες και υπεργρήγορη ευζωνική πρόσβαση. Σε ό,τι αφορά την ε, υπερφόρτωση, την ε, επιβάρυνση από το λεγόμενο ηλεκτροσμόκ, νομίζω ότι εδώ έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μεταφορά σημάτων από οπτικές σύνες που δεν είναι ηλεκτρομαγνητικά σήματα και αυτό μπορεί πραγματικά να βοηθήσει τη μείωση του ηλεκτρομαγνητικού σμόγκ το οποίο δημιουργείται και αυτό μας επιτρέπει με τις οπτικές σύνες να έχουμε ένα πυκνό δίκτυο το οποίο δεν δημιουργεί ακτινοβολία και επομένως επιβάρυνση για τον πληθυσμό. Και από την άποψη αυτή μπορούμε να κάνουμε μια τροποποίηση στο κείμενο για να ληφθούν υπόψη όλες αυτές οι παρατηρήσεις οι οποίες έχουν ε, διατυπωθεί σήμερα και νομίζω ότι έχουμε μια πολύ καλή συνένεση για τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακών Θεμάτων. Ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ Προθεσμοί για τροπολογιε ειναι είναι 24η Μαρτίου στι 12 το μεσημέρι, την επόμενη Πέμπτη δηλαδή. Όσοι, αυτοί, όσοι θέλουν να καταθέσουν τροπολογίε μπορούν ε, να τις καταθέσουν. Έχουμε δύο ακόμα γνωμοδοτήσεις. Ο Γιώκιμ Τσέλερ για τις προτεραιότητε σε ενεργειακή υποδομή και έχουμε τρεις σκιέ, τρεις σκιώδεις εισηγητέ. Σας συγκετεύω να σα δώσω τον πιο σύντομο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα κάνω κάθε προσπάθεια, γιατί είναι πάρα πολύ περίπλοκο το ζήτημα. Μιλάμε για την γνωμοδότηση για την Επιτροπή μας, για μία ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως και στην προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής, ε, μάλλον αρμόδια είναι η Επιτροπή Βιομηχανίας. Το θέμα είναι οι προτεραιότητες για την ενεργειακή υποδομή για το 2020 και μετέπειτα και ε, μια, ένα σύστημα για ένα νέο ευρωπαϊκό δίκτυο ενέργειας. το σύστημα της ενέργειας φυσικά είναι ιδιαίτερα επίκαιρο με τις πρόσφατες εξελίξεις. Είναι στενό το χρονικό πλαίσιο επειδή η Επιτροπή βιομηχανίας έκανε την ε, ακρόασή της και τη συζήτησή της και το Μάη ε, προβλέπεται η σχετική ψηφοφορία στην Επιτροπή προκειμένου μάλλον τον Απρίλιο θα πρέπει να ψηφίσουμε εμείς την γνωματοδοτησή μας. Αν θέλουμε εγκαίρως ε, να έχει η, Ευρωπα... η Επιτροπή βιομηχανίας την γνωματοδοτησή μας για το θέμα αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ περίπλοκο και πάρα πολύ σημαντικό. Για το ίδιο το θέμα τώρα, συζητώντας για την ενέργεια, καταλήγουμε γρήγορα στη στρατηγική το 2020. Μέχρι το 2020 το τμήμα των ανανεώσιμων ενεργειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ανέρχεται σε 20% στην παραγωγή ενέργειας. Θα πρέπει να μειωθούν 20% τα αέρια θερμοκηπίου. Υπάρχουν και κάποιοι αισιόδοξοι που μιλάνε για 30% μείωση εφόσον πληρούνται οι σχετικοί όροι και ενεργειακή αποδοτικότητα να αυξηθεί κατά 20% στα πλαίσια της εξοικονόμησης ενέργειας. Όλα είναι πολύ φιλόδοξα. Στόχοι, αλλά απέχουμε παρασφάγκες από αυτούς προς το παρόν. Και έχουμε ένα βασικό όρο όπου θα πρέπει να πετύχουμε την ανανέωση της υποδομής ε, της ενεργειακής, η οποία σε μεγάλο βαθμό είναι κακά συνδεδεμένη και επαπαλαιωμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία ε, ανέφερα, προβλέπει τρία σημεία. Μία ανάλυση της ε, τρέχουσας κατάστασης και αναφέρεται στις ανάγκες που προκύπτουν και ανακοινώνει τις πρωτοβουλίες που προτίθεται να αναλάβει προκειμένου στο θέμα των ενεργειακών υποδομών να πετύχουμε την ανανέωση των υποδομών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και έτσι προκύπτουν δύο μεγάλα θέματα. Το ένα είναι το θέμα της έγκρισης ε, σχεδίων και αυτό απασχολεί ιδιαίτερα την Επιτροπή μας γιατί τα θέματα έγκρισης πέρα από το ευρωπαϊκό επίπεδο αποφασίζονται σε εθνικό επίπεδο αλλά και περιφερειακό επίπεδο και κατά δεύτερον έχουμε και την χρηματοδότηση των σχεδίων και εδώ είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση. Οι χρηματοοικονομικές ε, ανάγκες, οι χρηματικές ανάγκες υπολογίζονται σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εξ αυτών μόνο τα μισά, οι μισές δαπάνες θα αφιερωθούν στην ε, ανανέωση των ενεργειακών υποδομών. Αυτά λοιπόν. Νομίζω ότι αυτές οι ανάγκες χρηματικές δεν θα μπορέσουν να καλυφθούν μόνο από την ε, πολιτική συνοχή και θα πρέπει να βρούμε την επόμενη ε, χρηματοοικονομική περίοδο πώς θα καλύψουμε τις υπόλοιπες ανάγκες να αυξηθούν τα μέσα. Θα πρέπει να αναζητηθούν λοιπόν νέε χρηματοπιστωτικέ ε, πηγέ. Και εδώ πέρα περιμένουμε προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό όμω που είναι απαραίτητο σε ό,τι αφορά τι πηγέ χρηματοδότηση είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει συντονισμό. Και επίση η ενεργειακή ενιαία αγορά θα πρέπει να αναβαθμιστεί, να συνεχίσει να εξελίσσεται. Επίσης, πολύ σημαντικό, το ανέφερα και προηγουμένως, αλλά το τονίζω εκ νέου, είναι η συμμετοχή του τοπικού και περιφερειακού επίπεδου και σε επίπεδο κρατών μελών σε ό,τι αφορά την έγκριση κατά το σχεδιασμό, μάλλον τον σχεδιασμό και την έγκριση νέων υποδομών. Ξέρουμε ότι όλοι είμαστε υπέρ της προστασίας του κλίματος, της εξοικονόμησης ενέργειας, της αλλαγής ε, και της μετάβασης σε εναλλακτικέ ε, πηγές ενέργειας, εφόσον φυσικά δεν ε, επηρεάζεται κανείς στο άμεσο περιβάλλον του. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις βλέπουμε ότι υπάρχουν έντονες αντιθέσεις και μεγάλη αντίσταση. Για παράδειγμα, αγρότες ε, στο Βραντεβούργο, οι οποίοι δεν θέλουν να μπουν ολικά πάρκα στη γειτονιά τους. και σε ό,τι αφορά την αποθήκευση άνθρακα. Θεωρούνται συχνά, θεωρείται συχνά ότι υποβιβάζεται το τοπίο, το περιβάλλον και είναι έντονες οι αντιθέσεις σε ό,τι αφορά και την ποιότητα ζωή συχνά ακούμε επιχειρήματα. Χρειαζόμαστε λοιπόν διαφάνεια στο σχεδιασμό αφενός σε όλα τα επίπεδα και μόνο αν υπάρξει πραγματική συνεργασία θεωρώ ότι πραγματικά αυτό αποτελεί αναπόσπαστη, αναπόσπαστο όρο θα μπορέσουμε να πετύχουμε τα σχέδιά μας αυτά και τους στόχους μας. Τώρα, για τι συστάσεις στην γνωματότηση, είχαμε κάποια επίσημα προβλήματα. Θέλαμε να περιοριστούμε στην γνωμοδότηση στα 1500-1500 χαρακτήρες. Να ευχαριστήσω τη γραμματεία της Επιτροπής και τον κύριο Καλέτα και την κύριο από την ε, ομάδα μου που καταφέραμε έστω και τμηματικά να αναφέρουμε σε έξι σημεία τα πιο σημαντικά θέματα. Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει η συζήτηση και ανυπομονώ να λάβω τις ε, σίγουρα πολλέ πολλές ε, τροπολογίες που θα λάβω για το θέμα αυτό. Θα προσπαθήσουμε με τους κοιότητες να τις διατυπώσουμε με τέτοιο τρόπο προκειμένου το θέμα της ε, πολιτικής της περιφερειακής σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό σχεδιασμό για την επόμενη δεκαετία να μπορέσει να συμβαδίσει. Uh, Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Έχω έξι υποψήφιους ε, ομιλητές, επτά. Και έχουμε ακόμα μία γνωμοδότηση για σήμερα. Ε, δεν βλέπω να έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε σήμερα την τελευταία γνωμοδότηση. Εκτός αν περιοριστείτε στο ένα λεπτό καθένας. Εν τη αυτή περίπτωση μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ξεκινάμε λοιπόν τη συζήτηση. Πρώτο η Μαρία Ιριγκογιάννη, η συγκήτρια, έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο τον πιο σύντομη. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Τσέλερ για την εργασία του, για το έγγραφο εργασία που μα έχει παρουσιάσει, που περιλαμβάνει την ουσία όλων αυτών των θεμάτων που θεωρώ και εγώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά για αυτό το ζήτημα. Νομίζω όμω ότι πρέπει να περιλάβουμε και μερικά ακόμα θέματα στην γνωμοδότηση αυτή τη Επιτροπή και να ενισχύσουμε περισσότερο ορισμένε ιδέε. πρέπει να αναφερθούμε στα γεωγραφικά προσκόμματα τα οποία αντιμετωπίσουν οι νησιωτικέ περιοχέ. Αυτό κάνει πολύ πιο δύσκολη την ενσωμάτωσή του στο ενεργειακό δίκτυο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό πρέπει να επιμείνουμε να υπάρξει μια κοινοτική στρατηγική η οποία να βασίζεται σε μεγαλύτερη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και την ε, πρόθεση των εναλλακτικών ενεργειών για να μπορέσουμε να μειώσουμε την ενεργειακή εξάρτηση αυτών των περιοχών από το εξωτερικό. Επίσης πρέπει να προωθήσουμε ευρωπαϊκού χαρακτήρα εργαλεία για την ενεργειακή υποστήριξη, κάτι το οποίο ξεκίνησε τον προηγούμενο χρόνο από την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να βοηθήσουν ορισμένε περιοχέ και πόλει. Τρίτον, πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση σε αυτά που λέει ο εισηγητή για τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και περιφερειών. Είναι απαραίτητο να υπογραμμίσουμε και να προωθήσουμε την περιφερειακή συνεργασία και το να τεθούν δεσμευτικοί στόχοι για τι διασυνδέσεις μεταξύ κρατών μελών, είτε μέσω ειδικευμένων περιφερειακών πλατφορμών, είτε μέσα από ιδιαίτερε πρωτοβουλίε. Τέταρτον, θεωρώ ότι μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο να ζητήσουμε από την Κομισιόν να είναι παρούσα και να υποβάλει μια πρόταση για τη δημιουργία ενός συστήματος αμοιβών και κινήτρων προς τις περιφέρειες ή προς τα κράτη-μέλη, ώστε να διευκολυνθεί όχι μονάχα η πιο γρήγορη διεκπαιρέωση των προγραμμάτων ευρωπαϊκού συμφέροντος, αλλά επίση και για την υποστήριξη τεχνολογικών επενδύσεων που θα οδηγήσουν σε σημαντικές βελτιώσεις τη ποιότητα ή την καινοτομία στα θέματα αυτά. Θέλω να ευχαριστήσω πάλι και τον κύριο Τσέλα για την εργασία του και θα παρουσιάσω ορισμένε τροπολογίε ακολουθώντα αυτά που είπε. Ευχαριστώ. Ε, και Μάνερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω το εισηγητή για έξοχη βάση που μας έδωσε Νομίζω ότι αξίζει να ενισχυθεί ο ρόλος της ε, πολιτικής συνοχής, κυρίως το πόσο, πώς χρηματοδοτούνται υποδομές ενέργειας, κυρίως αυτή την χρονική περίοδο, και λαμβάνοντας υπόψη το πόσο σημαντική είναι η στόχη της Ευρωπαϊκής Ενώσης του 2020. Η συνοχή σαφέστατα θα διδραματίσει σημαντικό ρόλο την επόμενη οικονομική περίοδο. Νομίζω ότι η παραγωγή ενέργεια σε τοπικό επίπεδο είναι ένα σημαντικό τομέα που δημιουργεί ευκαιρίες. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες σε διάφορους τομείς και πολύ συχνά μιλάμε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δυνατότητε παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας και αυτό πρέπει να αναφερθεί. Τρίτον, η ενεργειακή απόδοση. Το ανέφερε ο Γιωαχήμ όταν μίλησε. Νομίζω ότι αξίζει εδώ να υπογραμμιστεί ο ρόλος των ε, πόλεων και των μεγάλων αστικών κέντρων. Η αστική διάσταση στην περιφερειακή πολιτική είναι αξιοσημείωτη λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους για την ενεργειακή απόδοση. Τα διάφορα ξεχωριστά ταμεία κλπ. επικρίνονται εδώ Αυτά θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από τις μεγάλες ευρύτερε πολιτικές όπως η περιφερειακή πολιτική και η αγροτική. Ελίζα Πεθσουέντερ, λέει πρόεδρος. Äh, θα είμαι και εγώ πολύ σύντομη. Μου λείπει ένα κεντρικό σημείο σε αυτήν την ε, γνωμοδότηση. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λάβουμε υπόψη γιατί έχει να κάνει με την περιφερειακή προσέγγιση. Πρόκειται για το θέμα του πώς θα γίνει η κατανομή της χρηματοδότησης μεταξύ κεντρικών και αποκεντρωμένων δικτύων. Δεν πρόκειται λοιπόν μονάχα για μια χρηματοδότηση των ε, συγκεντρωτικών δικτύων. Αν θέλουμε τις αναπτυσσόμενες ανανεώσιμες ενέργειες να τις υποστηρίξουμε, θα πρέπει να βοηθήσουμε να υπάρχει και μια υποστήριξη των αποκεντρωμένων χώρων παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας που να συνδέονται με τα κεντρικά δίκτυα. Αυτό είναι λοιπόν μια μεγάλη διεκδίκηση που πρέπει να υποστηρίξουμε για τις ανανεώσιμες ενέργειες γιατί πρέπει ανάλογα με την περιοχή να έχουμε και διαφορετικές μορφές παραγωγής ενέργειας και φυσικά τίθεται και το θέμα της αποδίκευσης παραγόμενης ενέργειας. Πρόκειται λοιπόν το... Προκύπτει το ερώτημα αυτό και εμεί ω πράσινοι έχουμε προτείνει να γίνει μια τέτοια μελέτη από την Επιτροπή μας να δούμε πώς θα μπορέσουμε να συνδέσουμε τα αποκεντρωμένα δίκτυα με τα κεντρικά δίκτυα και ποια θα είναι τα αποτελέσματα τα οποία θα προκύψουν σε οικονομικό επίπεδο για τις περιφέρειες. Γι' αυτό ζητήσαμε να υπάρξει μια μελέτη και θα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το ποσοστό χρηματοδότηση των αποκεντρωμένων δικτύων. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να υπάρξει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια και για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω αυτών των δικτύων η, Καρ, η Καρμαντέλ. Ε, ευχαριστώ. Οι στόχοι της στρατηγικής του 2020 είναι και ο αγώνας κατά της, εν, της ένδυας. Αλλά υπάρχει μια νέα μορφή ένδυας που είναι η ενεργειακή ένδυα. Και αυτό αφορά τη στέγαση, τα κτίρια κτλ. Η μάχη για το κλίμα είναι και συγχρόνως μια μάχη για την σωστή απασχόληση. Αν έχουμε λοιπόν μια σωστή μόνωση των κτηρίων, αυτό θα δημιουργήσει και τοπικές θέσεις απασχολήσεω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης για τι χρηματοδοτήσει. Θα πρέπει να έχουμε μια μακροπρόθεσμη και όχι κοντόφθαλμη προσέγγιση, να, μην, να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Νομίζω ότι τα θέματα τη ενεργειακή απόδοση η Ευρώπη πρέπει να είναι φιλόδοξη και επομένω, ήδη από σήμερα, εγώ είχα κάνει μια πρόταση να δημιουργήσουμε ένα ειδικό ταμείο για την ενεργειακή απόδοση. Ας χρησιμοποιήσουμε λοιπόν την, ε, όλες τις ε, τράπεζες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη όπως είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και οι εθνικές όπως είναι η Καντεβέ στη Γερμανία κτλ. Για να επιτύχουμε το στόχο αυτό επίσης υπάρχει το θέμα των βελτίστων πρακτικών, κάτι το οποίο λείπει για τις ενεργειακές πρακτικές και επίσης ο κέριος ρόλος των πόλεων για το αν θα μπορέσουν οι πόλεις να έχουν μια άμεση χρηματοδότηση. Η άμεση σύνδεση μεταξύ των πόλεων και της χρηματοδότησης επομένω θα πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει Μπουστινάρου. Διακεκριμένοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να αναφερθώ στο θέμα που συζητάμε λέγοντάς σας Λοιπόν, για το θέμα που συζητάμε θα ήθελα να πω έχει υπάρχει ένα πρόβλημα τεχνικό ε, με το μικρόφωνο το μιλητή εντάξει έχει επιληθεί λοιπόν πάμε λοιπόν στις πρόσφατες δηλώσεις του Επιτρόπου Έτιγκερ πάνω απ' όλα υποδομές για κάποια χρονική περίοδο. Αυτό θα πρέπει να είναι ένα μέσο για να υλοποιήσουμε τους στόχους του 2020. Χρειάζεται υποδομή που είναι η υλική βάση για την ε, μετάδοση της ενέργειας. Δεύτερον, η υποδομή αποτελεί μια εναλλακτική για να αποφύγουμε την εξάρτηση από τη Ρωσία και για να αποφύγουμε διάφορες κρίσεις που μπορεί να παρουσιαστούν όπως βλέπετε τι γίνεται τώρα στη Βόρεια Αφρική, με την κρίση στη Βόρεια Αφρική. Η υποδομή μπορεί να είναι υπέρ του Ευρωπαίου καταναλωτή. Φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσει και λιγότερο για τις πολυεθνικές που ήδη έχουν τόσο μεγάλη επιρροή οι πολυεθνικές, ακόμα και στο Κοινοβούλιο. Μετά, κοινά κριτήρια για την ασφάλεια, για την εκμετάλλευση των πηγών και για να αποφευθούν καταστροφέ. Μη λησμονούμε την καταστροφή του κόλπου του Μεξικού και την καταστροφή στην Φουκουσίμα, στην Ιαπωνία. Όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο κείμενο. Ευχαριστώ, Ομπερ Μάιερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον συνάδελφο Τέλερ Να διευκρινίσω λίγο το δύο για την περιφερειακή στρατηγική ως ε, βάση των ε, διαμεθοριακών προγραμμάτων είναι κάπως ε, ασαφές. Θα έπρεπε να θέσουμε πιο συγκεκριμένα το στόχο και τη σύνδεση της στρατηγικής. Να συμπεριληφθούν συγκεκριμένες αναφορές. Γιατί στην πρακτική, στην πράξη, είναι σημαντική και η στρατηγική για το Δούναβη και θα πρέπει να λάβει συγκεκριμένα ε, ζητήματα και σε ό,τι αφορά διαμεθοριακά προγράμματα, σε ό,τι αφορά και τις παλιές τεχνολογίες, ε, τις πυρηνικές τεχνολογίες και είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παρουσιάσει κάτι. Νομίζω λοιπόν ότι έχει απευθυνθεί έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι' αυτό λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση θα υποβάλω σχετικές τροπολογίες να μην είναι μόνο αφηρημένη η διατύπωση, το οποίο καλό είναι και αυτό, αλλά να έχουμε και συγκεκριμένες προτάσεις. Ο Τζιβλάσακ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ένα-δύο πράγματα σχετικά με το θέμα που συζητούμε. Αναφερόμαστε στις υποδομές της ενέργειας και δεν πρέπει να ξεχνάμε και την χωροταξία και δεσυνοριακό συντονισμό τέτοιων προγραμμάτων χωροταξικών. Η βασική παράμετρος, οι βασικοί παράμετροι για την ενεργειακή απόδοση αναφέρθηκαν. Δηλαδή, χρειαζόμαστε καλύτερο δίκτυο, το οποίο θα έχει λιγότερες απόδο, ε, όσον αφορά την ενέργεια. Επιπλέον, η διαδικασία του σχεδιασμού, οι κανόνες για το σχεδιασμό και η χορήγηση των αδειών. Όλα αυτά θα πρέπει να καλυφθούν διαφορετικά ίσως οι κανόνες για, την, για το σχεδιασμό, ίσως να εμποδίσουν τα μεγάλα έργα. Πολύ σύντομα, πολλά υπόθηκαν για την ανανεώσιμη ενέργεια κλπ. Και συμφωνώ με αυτά που υπόθηκαν. Όσο περισσότερε τι πηγέ, τόσο καλύτερα. Κυρίω φυσικέ καταστροφέ που ζήσαν πρόσφατα και στην Ιαπωνία το δείχνουν αυτό. Και προβλήματα, η κρίση στη Βόρεια Αφρική κλπ. Και εμεί πρέπει στην πατρίδα μα, στην περιοχή μα, να είμαστε αποδοτικοί, όσο πιο αποδοτικοί γίνεται. Για την ενεργειακή απόδοση δεν ε, έχουμε το υπογραμμίσει όσο χρειάζεται το θέμα. Διάβασα με ενδιαφέρον το έγγραφο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χρειάζεται να κινηθούμε πολύ πιο γρήγορα πάνω σε αυτό το θέμα. Θα πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση, οι εθνικές αρχές να τα καταφέρουν πολύ καλύτερα στον αφορά του σχετικού στόχου. Για τα δημόσια κτίρια, τα ιδιωτικά κτίρια, τα νέα κτίρια, τι μεταφορές, του δρόμους και τι συσκευέ κάθε είδου. Τεράστιο πεδίο, τεράστιο περιθώριο για βελτιώσει. Και είναι εξίσου σημαντικό λοιπόν να το τονίσουμε και αυτό όσο και να τονίσουμε και τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Ευχαριστώ, Ιωαχήμ. Μισό λεπτό εσύ το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να σα ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τι πολύτιμε συνεισφορέ σα. 1500 χαρακτήρε. είναι το όριό μα. Επομένω, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομο. Κυρία Σουέντερ, προφανώ και και εμένα είναι δική μου μέρημνα ότι δεν πρέπει τα κεντρικά δίκτυα να χρηματοδοτούνται από περιφερειακά κονδύλια. Η Κομισιόν από την άλλη πλευρά έχει ζητήσει να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ των υποδομών προτεραιοτήτων για την ευρωπαϊκή διασύνδεση ενεργειακών πηγών και χωριστά αυτά που έχουν να κάνουν με τις περιφέρειες. Και υπάρχουν οι περιοχές που έχουν προβλήματα λόγω γεωγραφικής θέσης, υπάρχουν άλλες περιοχές που έχουν ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες, ήλιο και άνεμο λοιπά Και εκεί μπορεί πράγματι να εξασφαλιστεί η απεξάρτησή τους από εισαγόμενο πετρέλαιο και ορυκτές πηγές. Ακολουθώντας το, δρόμο αυτό είχα μονάχα αυτό το μισό λεπτό και δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο παρά ο μονάχα ότι χαίρομαι για όλα αυτά τα οποία ακούσατε και περιμένω να δω και τις τροπολογίες σας και θα έρθω σε επαφή με τους σχεδόντες συζητητές για την τελική διαμόρφωση της νομοδότησης. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ιωχήμ. Λοιπόν, 24 Μαρτίου στι 12 είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Την 5η, 12 το μεσημέρι, η προθεσμία τροπολογή έκθεση του κ. Τσακίρσκη όσον αφορά την κοινή αγροτική πολιτική. Θα ήθελα λοιπόν όσοι θέλουν να πάρουν το λόγο να μας το πούν τώρα, ώστε να μπορέσουμε να δούμε πόσο χρόνο έχει ο καθένας. Λοιπόν, στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την κοινή αγροτική πολιτική και το ποια προσέγγιση ακολουθηθεί μέχρι το 2020, λοιπόν αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε και όσον αφορά σαν πρόβλημα όσον αφορά την χορήγηση τροφίμων και την χρήση των φυσικών πόρων. Με άλλα λόγια είναι ένα θέμα το οποίο ξεπερνά την παραδοσιακή προσέγγιση της κοινή αγροτικής πολιτικής. Η κοινή αγροτική πολιτική η οποία είχε συμπεριληφθεί σε θήκη της έρευνας αναφέρεται στην γενική πρόσβαση στα τρόφιμα σε προσβάσιμες τιμές και αξιοπρεπές εισόδημα για τους ε, γεωργούς. Με άλλα λόγια αναφέρεται στην ασφάλεια των τροφίμων, στην ποιότητα των τροφίμων, στην πρόσβαση στις προδιαγραφές για τα τρόφιμα η κοινή αγροτική πολιτική ε, πέρασε μια διαδικασία επαναστατικών αλλαγών. Η ΚΑΠ είναι περίπου το 40% του προϋπολογισμού και η πολιτική της συνοχής έχει ξεπεράσει ε, την κοινή αγροτική πολιτική όσον αφορά το ποσοστό του προϋπολογισμού που καταναλώνει. Λοιπόν, η κοινή αγροτική πολιτική εδράζεται επί της αρχής των άμεσων πληρωμών και η γεωργία όλο και περισσότερο ε, υπόκειται στους κανόνες της αγοράς. Ε, γινόταν πάρα, πολύ, πάρα πολλές αναποτελεσματικές παρεμβάσεις στην αγροτική πολιτική ε, και ήταν και πολύ δαπανηρές. Πολύ συχνά παραβιάζονται στους κανόνες του ΠΟΕ. Ο χαρακτήρας της παρέμβασης πρέπει να εξετάζεται. Πόσο σημαντική είναι η παρέμβαση για τον τομέα. Ποια είναι η φύση της, ποιο είναι το κόστος, κόστος της παρέμβασης. Θα ήθελα να αναφερθώ γενικά στους Ευρωπαίους γεωργούς η γεωργοί λοιπόν της Ευρώπης παίρνουν το 55 με 60% του εισοδήματος εκείνων που ζουν και εργάζονται μάλλον σε άλλους τομείς. Ένα σημαντικό κομμάτι αυτού αποτελείται από επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ισχύει για τους γεωργούς και στα παλιά και στα νέα κράτη-μέλη. Φεύγουν από τη γη, από την Ήπεθρο, οι γεωργοί, φεύγουν οι νέοι γεωργοί, γυράς και ο πληθυσμό και χειρότερο απ' όλα. Η ζωή πεθαίνει σε πολλά σημεία της Ήπεθρου. Σβήνει. Η γεωργία ε, δεν είναι κάτι που αφορά μόνο την γεωργική παραγωγή, αφορά την παραγωγή διαφορών ε, δημοσίων αγαθών. Κάποια από αυτά τα αγαθά ε, δεν πληρώθηκαν δεόντως, δεν αποζημιώθηκαν σωστά για τους κόπους τους οι γεωργοί κατά παρελθόν. Έγινε ο υγείας της κοινή ερωτικής πολιτικής το 2008. Και εκεί, σε αυτόν τον απολογισμό, έγιναν κάποιες διαπιστώσεις, ε, κάποιες αναποτελεσματικότητες όσον αφορά την ΚΑΠ και η έκθεση έδειξε ποια θα πρέπει να είναι η πορεία της ΚΑΠ στο μέλλον, τα πορίσματά της, τα πορίσματα του απολογισμού. Το Νοέμβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μια έκθεση. Θέμα της έκθεσης το μέλλον της κοινή αγροτικής πολιτικής η Επιτροπή Γεωργίας, ο κύριος Ντες, ο Ευρωβουλευτής, ο κύριος Ντες, ε, συντάσσει μια έκθεση. Η γνωμοδότησή μου είναι πολύ σύντομη και βασίζεται επί της απόψεως της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το, στο πρώτο σημείο αναφέρονται οι βασικές προκλήσεις για την κοινή αγροτική πολιτική Κάποιοι από εσά ίσως ε, να έμειναν έκπληκτοι διότι αναφέρομαι στην κοινή ερωτική πολιτική σαν κινητήρα ανάπτυξη. Την τελευταία 20 ετία εμεί είδαμε αποτελμάτιση όσον αφορά την γεωργική παραγωγή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ σε άλλε περιοχέ του κόσμου είχαμε αύξηση μέχρι 200% όσον αφορά την παραγωγικότητα. Άρα λέω ότι πρέπει να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας στη διεθνή αγορά μέσω της ΚΑΠ. Θα πρέπει τα μέτρα να έχουν σαν στόχο την αγορά, να λαμβάνουν υπόψη την παραγωγή των δημοσίων αγαθών που παράγουν οι γεωργοί. Αυτό συμπεριλαμβάνει την ασφάλεια των τροφίμων, την διατήρηση της βιοπικιλότητας, τη σωστή διαχείριση των δασών και των υδάτων, γιατί είναι σημαντικό κομμάτι των γεωργικών δραστηριοτήτων. Και μετά βιώσιμη ανάπτυξη η οποία θα βασίζεται επί της γνώσεως και επί της εκπαιδεύσεως. Με άλλα λόγια, αυτά τα οποία έχει στερνιστεί η στρατηγική για το 2020. Όλα αυτά θα βελτιώσουν τη συνοχή. Οικονομική συνοχή, κοινωνική συνοχή, περιβαλλοντική συνοχή κλπ. Στην παράγραφο 2 αναφέρομαι στις ε, διαφορές που υπάρχουν στον αγροτικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Οι άμεσες πληρωμές βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα και τα εισοδήματα των εκμεταλλεύσεων και συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και βοηθάνε στο να διατηρηθεί το δυναμικό του εδάφους. Επίσης, αναφέρομαι στα αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την άμεση στήριξη. Και υπάρχει ανάγκη να απομακρυνθούμε από τις ημερομηνίε αναφοράς που χρησιμοποιούμε τώρα, τις περιόδους αναφοράς, γιατί είναι πολύ απόμακρες στο παρελθόν. Στην επόμενη παράγραφο Αναφέρομαι στην ποικιλομορφία του μεγέθου των εκμεταλλεύσεων, τι διαφορέ που υπάρχουν όσον αφορά τα μεγέθη των εκμεταλλεύσεων. Οι μικρέ οικογενειακέ εκμεταλλεύσει δημιουργούν απασχόληση, δίνουν δουλειά στον κόσμο, ε, προστατεύουν την απασχόληση και δημιουργούν αυτά τα δημόσια τα αγαθά. Λέω ότι χρειάζεται να διατηρηθεί η ποικιλομορφία των μεγεθών των εκμεταλλεύσεων στην Ήπεθρο, διότι αυτό διαφυλάσσει το μέλλον του ευρωπαϊκού αγροτικού μοντέλου, θα διατηρήσει την παραγωγή σε λογική κλίμακα και αυτό είναι κάτι που βελτιώνει την ποιότητα και τη γεύση των αγροτικών προϊόντων. Στην παράγραφο 4 λέω ότι η ύπεθρος και η γεωργία δεν αφορούν μόνο τη γεωργική παραγωγή αλλά την παραγωγή πόρων για τη βιομηχανία, την παραγωγή ανανεωσίμων πόρων και είναι και είναι, υπάρχουν η δυνατότητα για ανάπτυξη πέθρου, του τουρισμού κλπ, πολιτισμικά χαρακτηριστικά, ε, πολιτισμική κληρονομιά όπως ε, διάφορες συνταγές, ε, διατροφικές παραδόσεις κλπ. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, σημαντικές πτυχές ε, της περιφερειακής ανάπτυξης. Στην τελευταία παράγραφο αναφέρομαι στην ανάγκη να διατηρηθούν τα κοινοτικά κριτήρια για την κατανομή χρηματοδοτήσεως ε, στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα. Δεύτερος πυλώνας αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου. Οι υποδομές για την ανάπτυξη της υπαίθρου και τεχνικές υποδομές και υποδομές από πλευράς κοινωνικής και παιδεία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να παραμείνει ζωντανή ύπεθρο. Και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό ο δεύτερος πυλώνας να έχει έναν ευρύτερο ρόλο να διαδραματίσει από αυτόν που περιγράφεται στην έκθεση DES. Η έκθεση DES αναφέρεται στο πρασίνισμα του δεύτερου πυλώνα. Οι περιβαλλοντικές πτυχές είναι βέβαια σημαντικές, αλλά θα πρέπει να υπογραμμίσουμε περισσότερα στοιχεία για την ανάπτυξη πέθρου πέρα από το περιβάλλον. Πρέπει να μιλάμε και για την ανάπτυξη της υπαίθρου που ξεπερνά τις γεωργικές πτυχές και τις πτυχές του, του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να αφορά η ανάπτυξη της υπαίθρου και ένα ευρύ φάσμα άλλων πτυχών συναφών. Υπάρχει η ανάγκη συντονισμού. Χρειάζεται κάτι τέτοιο. Χρειάζεται συντονισμός μεταξύ των τεσσάρων πέντε επιτρόπων που είναι υπεύθυνοι. Χρειάζεται όμως ο συντονισμός διότι άνευ αυτού δεν μπορείς να εκμεταλλευτεί πλήρω την πολιτική συνοχή ή την κοινή αγροτική πολιτική, που είναι πάρα πολύ σημαντικέ πολιτικέ. Θα πρέπει να κινηθούν μαζί για να αναπτυχθεί η ύπεθρο οι δύο Λοιπόν, παρα... ο, ο Λουί Άλβε έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θέλω να χαιρετήσω το έργο του κυρίου Σικέρσκη για όλα αυτά τα θέματα, όπου είναι πολύ σημαντική και η γνωμοδότησή μα, παρά το γεγονό ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ σύντομη και θα ήθελα να παρουσιάσω τη θέση της Σοσιαλιστικής Ομάδας για τα θέματα αυτά. Η γεωργική πολιτική στον ορίζοντα του 2020 θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις ό,τι αφορά τα τρόφιμα, του φυσικούς πόρους, αλλά και τις εδαφικές προκλήσεις. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να έχουμε στόχους, στόχους βιώσιμους για την παροχή των τροφίμων και να είναι και ανταγωνιστική συγχρόνως, μια βιώσιμη ε, προστασία των ε, ε, διαθέσιμων πόρων για να αποφύγουμε και την αλλαγή λόγω κλιματικής αλλαγής και επίσης να εξασφαλίσουμε και μία ισορροπία σε επίπεδο εδαφικό και νομιμοποίηση και αποτελεσματικότητα και ισοδίκαια κατανομή των πόρων στα κάτι μέλη. Πρέπει να ξεπεράσουμε τα ιστορικά κριτήρια και να διανύμουμε με ισοδίκαιο τρόπο τα ποσά στις ε, χώρες και στους γεωργούς και επίση να εξασφαλίσουμε και μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των προϊόντων που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτών τα οποία παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι σημαντικό και για να εξασφαλίσουμε του παραγωγού εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να έχουμε μια πολιτική λοιπόν η οποία θα επιτρέψει στη γεωργία σε όλε τι περιοχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρηθεί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό υπό την έποψη τη περιφερειακή πολιτική. Θα πρέπει λοιπόν η κατανομή των πόρων του δευτέρου πυλώνα να λάβει υπόψη και στοιχεία εδαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης η κοινή αγροτική πολιτική δεν πρέπει να αφήσει την αγορά να λειτουργεί από μόνη της, θα πρέπει να έχει τη δική της κυριαρχία για τα θέματα αυτά και θα πρέπει να υπάρξει και μια διαχείριση κινδύνου για την γεωργία, όπου και οι αγροτικές ασφαλίσεις παίζουν ένα ιδιαίτερο ρόλο. Χρειαζόμαστε να υπάρχει ανανέωση των περιοχών που είναι ακριτικές και νησιωτικές, δημιουργία θέσεων απασχόλησης, να δημιουργηθούν οι μηχανισμοί οι οποίοι θα δώσουν στους νέους τα κίνητρα να παραμείνουν στις περιοχές αυτές τις αγροτικές, όχι μόνο στη γεωργία, αλλά για την παραγωγή υπηρεσιών οι οποίες είναι ειδικευμένε είτε προς την κατεύθυνση της γεωργίας είτε άλλε υπηρεσίες οι οποίες βοηθούν την αγροτική οικονομία και με τον τρόπο αυτό να δώσουν μεγαλύτερο δυναμισμό και να εξασφαλίσουν και μια μεγαλύτερη <clears throat> ε, δραστηριότητα στον αγροτικό χώρο που είναι απαραίτητη για να παραμείνει ο πληθυσμός στις περιοχές αυτές. Αυτά προς το παρόν θα ήθελα να αναφέρω ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Σικέρσκι για την γνωμοδότηση που ετοίμασε. Πολύ σύντομα θα ήθελα να επενθυμίσω κάποια στοιχεία που κατά την άποψή μου είναι πάρα πολύ σημαντικά. Εφόσον μιλάμε για το μέλλον της κοινή αγροτικής πολιτικής, η προσαρμογή του συστήματος των πόρων, των γεωργικών ταμείων και τα κριτήρια που θα χρησιμοποιούνται για τις άμεσες πληρωμές στη Γεωργία ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Γιώργος. Άλλο στοιχείο είναι η βελτίωση ε, των συμβουλών που παρέχονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Για του γεωργού. οι συμβουλέ βοηθούν του γεωργού, να αξιολογήσουν τι επιδόσεις του, τι επιδόσει τη εκμετάλλευσής του και συνεπώ με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν οι γεωργοί να καταρτήσουν, να αποφασίσουν προτεραιότητε. Άλλη πτυχή πάρα πολύ σημαντική κατά την άποψή μου, κάτι που ανέφερε και ο Σικέρσκι, Δηλαδή ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε τα κριτήρια της συνοχής και να βελτιώσουμε το συντονισμό μεταξύ της κοινής αγροτικής πολιτικής και της πολιτικής περιφερειακής συνοχής. Μιλήσαμε και για την πολιτική περιβάλλοντος. Έχει σημασία και η προστασία του περιβάλλοντος. Χρειάζεται ισορροπία μεταξύ των πτυχών των περιβαλλοντικών και της αναπτύξεως της υπαίθρου, ούτως ώστε όλα αυτά να γίνουν προς όφελος όλων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Μάνες. Θέλω να πω κάτι σε σχέση με το, τα θέματα που αφορούν τους ε, <clears throat> εργαζόμενους στον αγροτικό τομέα. ήδη στη χώρα μου, στην Φιλανδία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μέτρο χιόνι ή δύο. Και χρειαζόμαστε λοιπόν να έχουμε μια πολύ, ένα πολύ ισχυρό δεύτερο πυλώνα, τον πυλώνα της αγροτικής ανάπτυξης δηλαδή, και επομένως είναι απαραίτητος ο ρόλος της χρηματοδότησης στα θέματα αυτά, ώστε τα μέτρα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη να βρίσκονται όλα στο δεύτερο πυλώνα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και το ρόλο των δασών και τα δάση βρίσκονται μέσα στην κοινή αγροτική πολιτική και εμείς έχουμε τονίσει στο παρελθόν πόσο σημαντικά είναι τα θέματα της εκμετάλλευσης από οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, λέει ο κύριος Βλάσακ. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σικέρσκι για αυτή την πάρα πολύ ευρία γνωμοδότηση, την δέχομαι θετικά. Υπογραμμίζει σωστά την όλη η προβληματική, την εδαφική και τη σημασία που έχει ο δεύτερος πυλώνα τη κοινή αγροτική πολιτική. Και εγώ πιστεύω ότι για να μην έχουμε αρνητικές συνέπειες όσον αφορά την Υπέθρο. θα πρέπει να ενισχύσουμε τις υποδομές, τις υπηρεσίες και να εγγυηθούμε αρκετές θέσεις εργασίας στον τομέα της Υπέθρου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τσέστα, θες να πεις κάτι? Ένα λεπτάκι μόνο. Συμφωνώ με τις απόψεις των συναδέλφων και τη συμπεριέλαβα στην γνωμοδότηση που αρχικά είχα καταρτήσει, αλλά δυστυχώ έπρεπε να περιοριστεί σε έκταση. Η ΚΑΠ θα πρέπει να προσαρμοστεί από περιφερειακή οπτική γωνία. Επίση, συμφωνώ με τη μεταφορά καινοτομία και τεχνογνωσίας. Το 2050 θα έχουμε 9 δις ε, κατοίκους ε, στον κόσμο και θα πρέπει να παράγουμε 80% πιο πολλά τρόφιμα στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη 40 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε φτώχεια, σε συνθήκες φτώχειας. Αυτά τα προβλήματα είναι σοβαρά. Και αν υπομονώ να λάβω τα σχόλια των συναντέλφων και φυσικά όλα θα συμπεριληφθούν στην γνωμοδότηση. Η Πρόεδρος, όπως και στις άλλες τροπολογίες, 24 Μαρτίου, 12 η ώρα το μεσημέρι είναι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών για όσους θέλουν να καταθέσουν τροπολογίες. Και έτσι θα λήξει η σημερινή μας συνεδρίαση. Τώρα έχουμε συνεδρίαση των συντονιστών. Αύριο το πρωί στις 9 λοιπόν θα τα πούμε. Έχουμε πολλές ψηφοφορίες. Μην ξεχάσετε τις κάρτες σας. Ευχαριστώ και παρακαλώ να <laughs> φύγετε γρήγορα και ήσυχα προκειμένου να ξεκινήσουν τη συνεδρίαση τους οι συντονιστές.